Dear colleagues, please, may Συνάδελφοι, ξεκινάμε. First with the adoption of the agenda. May we consider it adopted. Thank you. Θεωρείται δεκτή η μερισία διάταξη. Έχω να κάνω κάποιες ανακοινώσεις επίσης. Όπως γνωρίζετε, σήμερα έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος από τις φρικτές τρομοκρατικές επιθέσεις της Βρυξέλλες. Στις 10 λοιπόν πρέπει να πάμε μπροστά από το ημικύκλιο. Θα διακόψουμε λοιπόν τη συνεδρίασή μας στις 9.55 για 10 λεπτά. και στις 10 και 5 θα επανέλθουμε. Τώρα συστάσεις και αποφάσεις από τους συντονιστές χθες. Συμφωνήθηκαν τα εξής. Να στείλουμε μία επιστολή στο CCC λέγοντας ότι όλες οι εκθέσεις αυτές είναι εκτός ποσοστώσεων και θα πρέπει να κατατεθούν οι προτάσεις ε, μέχρι τις 24 Μαρτίου το μεσημέρι. Το Action Plan για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Ενίσχυση των εθνικών αρχών για τον ανταγωνισμό, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ε, Τραπεζική Ένωση ECR, η ALDE, σύμφωνα με την πολιτική εναλλαγή, θα ενδιαφερθεί για την έκθεση αυτή του χρόνου ετήσια έκθεση ALDE για τον ανταγωνισμό, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Σοσιαλδημοκρατητές, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες Σοσιαλιστές, γνωμοδότηση για την αλλαγή στους μεταρρύθμιση στους ιδίους πόρους ε, ε, σοσιαλιστές, εφαρμοστικές ε, εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από το Προεδρείο, έλεγχος εφαρμοστικών πράξεων για τα κρύψ Θα υπάρξει ψηφοφορία στις 27 Μαρτίου, κατάθεση τροπολογιών μέχρι τις 23 Μαρτίου. Το Μάιο θα εξετάσουμε τα θέματα των των εταιριών βαθμολόγησης και αξιολόγησης. Θα συναντηθούμε με τον Ινιάσιο Βίσκο της Ιταλικής Κεντρικής Τράπεζας για τα CCTB και CCTB έχει εγκριθεί το πρόγραμμα. Οικονομικός διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο για τις ειδικέ ανακράτως εκθέσεις θα οργανωθεί στις 30 Μαΐου. Και τέλος, δύο μέλη της ΕΚΟΝ, Μάντο και Μορέλ, θα πάρουν μέρος στο δίκτυο αναφορών. Περνάμε στο πρώτο θέμα λοιπόν, το τέσσερα δηλαδή. Μια πολύ σημαντική νομίζω ακρόαση για την εξυγίανση και την ανάκαμψη των αντισυμβαλωμένων κεντρικών αντισυμβαλωμένων μετά από την οικονομική κρίση αναγνωρίστηκε ο κεντρικός ρόλος των ε, κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Έχουν ε, μετά τις αποφάσεις που έχουμε πάρει περισσότερες, δώσει περισσότερες αποστολές, καθήκοντα, στους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους υπόκεινται σε αυξημένο έλεγχο σε σχέση με το παρελθόν και είναι πλέον συστημικά σημαντικά όργανα. Ταυτόχρονα έχει υπάρξει πρόοδος για τη διαχείριση κινδύνου και την καθημερινή διαχείριση των CCP, το PRT επίσης έχει εφαρμόσει μέτρα για τον έλεγχο ε, των μελών clearing των CCP. Επίσης ε, ε, δεν αποκλείουμε την εξέταση σεναρίων τα οποία προβλέπουν ότι ένας κεντρικός αντισυμβαλόμενος έχει να αντιμετωπίσει υψηλού επίπεδου κρίσης, σοκ κάτι το οποίο εμπλέκει υποχρεωτικά και τις εθνικές αρχές ε, για την ε, ανάκαμψη και την εξυγίανση. Έχουμε υιοθετήσει σαν έκθεση, μία έκθεση το 2013 ε, για το πλαίσιο των διαδικασιών εξυγίανσης. Η πρόταση την οποία έχουμε μπροστά μας νομίζω ότι προβλέπει μέσα και κίνητρα για την πρόληψη των κρίσεων και την σωστή τους διαχείριση αν πράγματι υπάρξουν κρίσεις. Δείχνει ποια είναι η κατάσταση των συζητήσεων σε διεθνές επίπεδο Ε, υπάρχουν ε, οργανισμοί που ασχολούνται ειδικά με την ανάκαμψη, όπως επίσης και ειδικότερα με την εξυγίανση των αντισυμβαλωμένων και γι' αυτό ακριβώς ε, νομίζω στα πλαίσια αυτού του περίπλοκου θέματος έχουμε πολύ σημαντικούς εκπροσώπους. Έχουμε την Έλκε Κένινγκ, την πρόεδρο της SRB, όπως επίσης και της ομάδας εργασίας για την εξυγίανση Έχουμε τον Στίβεν Μαϊτζούρ, ο οποίος θα μας μιλήσει για την αγορά των παραγόγων. Εμείς σαν συνομοθέτες προσπαθούμε να δούμε ποια είναι τα συμφέροντα των κεντρικών αντισυμβαλωμένων χωρίς να θίξουμε κανέναν άλλον από τους εμπλεκομένους. Γι' αυτό θα έχουμε στο δεύτερο πάνελ τον Έρικ Müller που εκπροσωπεί τα CCP, το Eurex Clearing, ο Μακόρμικ, ο οποίος ε, εκπροσωπεί μια διαφορετική εταιρεία και την Κέρι, η οποία είναι υπεύθυνη για ανάλυση κινδύνου στο BlackRock, στην BlackRock. 7 με 8 λεπτά ο καθένας παρακαλώ για να κάνετε τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Μετά θα υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής. Έχετε 3 λεπτά για τις ερωτήσεις σας και 3 λεπτά και οι ε, προσκεκλημένοι μας για να απαντήσουν. Θα δώσω στο τέλος τον λόγο στην Κέιτ Σουίμπορν και τον Ιάκομ Φον Βάιτσέκερ για τις καταληκτικές τους παρατηρήσεις. Θέλω να καλωσορίσω την Έλκο Κένιν και της δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε για να σας μιλήσω για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Για μια πολύ, μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα για την Ευρώπη και για τις Βρυξέλλες. Να σα εξηγήσω καταρχά, γιατί υπάρχει τόσο ενδιαφέρον για τους CCP, για του κεντρικού αντισυμβαλόμενους. Οι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι αποτελούν ε, ακροκονία όλοι για τις μεταρρυθμίσεις μετά την κρίση στις ε, αγορές, στι εξωχρηματιστριακές, γιατί μειώνουν τον κίνδυνο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αλληλοσύνθεση των μεγάλων τραπεζών και παράλληλα αυτό είναι μια ωραία εικόνα οι CCPs θα πρέπει να είναι στεναροί και αυτό συνεπάγεται και κάποια διαχείριση κινδύνου, ε, stress test και πολλά από αυτά έχουν ήδη ξεκινήσει και περιλαμβάνει και αυτό λείπει τώρα την ανάκαμψη και την εξυγίανση σχέδια τέτοια για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους. Η SRP ως η αρχή εξυγίανσης ε, έχει τέτοιο ενδιαφέρον για να καθορίσει ένα πλαίσιο εξυγίανσης για το CCPs. Γιατί κυρίως οι μεγάλες τράπεζες είναι μέσα εξυγίανσης των CCP. Όχι μόνο αυτές ε, στην που είναι στην Ευρωζώνη. Και γι' αυτό εκτίθενται στον κίνδυνο των συνεπαγόμενων των CCP. Άρα, αν υπάρξει κίνδυνος για τα CCP, αυτό θα επηρεάσει και τα μέλη εξυγίανσης και α, το αντίστροφο ισχύει επίσης ε, για τη μεγάλη αποτυχία του CCP κατά πάσα πιθανότητα ε, σημαίνει αποτυχία ενό ή περισσότερων μέλων, μέλων Και γι' αυτό λοιπόν παρακολουθούμε στενά τα, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θέμα αυτό και όπως είπατε ενεργά συμμετέχουμε και στην ε, εργασίες του Συμβουλίου Χρηματοστατικής Σταθερότητα και σε ό,τι αφορά την εξηγήση των CCP και σε ό,τι αφορά τις αλληλεπιδράσει μεταξύ CCP και οι τελευταίοι ε, καταθυντήρες γραμμές ε, που καταρτίστηκαν από την Επιτροπή της οποίας προεδρεύω στο ΣΟΣΠΗ αναμένεται το καλοκαίρι του 2017. Τώρα, γιατί βρισκόμαστε εδώ. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σχέδιο εξυγένσης και ανάκαμψη του CCP που δημοσιεύτηκε το Νοέμβριο, το οποίο συνάντησε γενικέ γενικές γραμμές με τι διεθνεί εξελίξει, εμεί ω ε, SRB καλωσορίζουμε την πρόταση αυτή και καλωσορίζουμε το γεγονό ότι εξασφαλίζει στις ότι οι αρχέ ε, εξηγήνση τραπεζών, συμπεριλαμβανομένες και τη SRB, θα συμμετέχουν στη διαδικασία ω παρατηρητέ. στη νέα Επιτροπή Εξυγίανσης ε, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών της ΕΣΜΑ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ των ε, αρχών να συντονίζεται, να είναι οργανωμένη και θα πρέπει λοιπόν αυτό να αφορά όχι μόνο τις αρχές που θα πρέπει να συμμετέχουν στο σώμα εξυγίανσης, αλλά να υπάρχει και μία υποχρεωτική διαμεσολάβηση σε περίπτωση διαφωνίας. Και να σας πω ότι διεθνώς υπάρχει και δέσμευση να σχηματιστεί να σχηματιστούν ομάδες διαχείρισης κρίσεων για τους μεγάλους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους ΕΣΥΠΗΣ. Φυσικά όλα επιδέχονται βελτίωση. Υπάρχουν λοιπόν τρεις τομείς όπου θα μπορούσαμε να εκφράσουμε και άλλες σκέψεις. Ο πρώτος τομέας στον οποίο θα ήθελα να επικεντρωθώ είναι το πώς μεταχειριζόμαστε τα μέλη εξυγένσης. Σε περίπτωση αποτυχίας ενός μέλους ε, εξυγένσης, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποτυχία του CCP. Και τότε λοιπόν, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να δούμε πώς το CCP μπορεί να βοηθηθεί, αλλά αυτό που ουσιαστικά γίνεται είναι ότι επιβάλλονται απώλειε στα μέλη εξυγίανση σε, σε μια φάση που ενδεχομένω να υπόκειται ήδη πιέσει. Άρα, η εξυγίανση των μέρων, των κεντρικών αντισυμβαλωμένων, δεν ε, α, καταδεικνύει ότι ο κίνδυνος αλληλεπίδρασης έχει μεταφερθεί. Δεν είναι μόνο θέμα μεταξύ τραπεζών, αλλά και μεταξύ κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Και το πρόβλημα, όπω σα είπα, ανακύπτει ιδιαίτερω αν η εξυγίανση μια τράπεζα δεν μπορεί να γίνει επιτυχώ. Για παράδειγμα, λόγω α, έλλειψης ε, τέτοιων ευθυνών. Άρα υπάρχει ε, μια εξάρτηση από την επιτυχή εξυγίανση των τραπεζών. Είναι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος ουσιαστικά. Και γι' αυτό λοιπόν ίσως θα χρειαζόταν waiver για κάποιες υποχρεώσεις, για κάποια μέλη. Για παράδειγμα, να υπάρχει απαλλαγή από πρόσθετες θέσεις για τα μέλη εξυγένσης που είναι ήδη υπό εξυγένσης ή σε περίπτωση που υπάρχει ε, περίπτωση απορρόφησης των ε, απολειών. Και πάλι για μέλη που έχουν, είναι ήδη υποπίεση. Δεν υπάρχουν φυσικά θαύματα, δεν μπορούμε να αποφύγουμε εντελώς τις απώλειες, άρα ενδεχομένως να χρειαστεί να υποστούν μεγαλύτερο ποσοστό απώλειων ή ενδεχομένως να χρειαστεί να κατανεμηθούν και σε έμεσα μέλη εξυγίανσης ή απώλειες, τα οποία ως τώρα ενδεχομένως δεν ήταν σε κίνδυνο. Ένα δεύτερο θέμα που ήθελα να αφήξω για να ξεκαθαρίσω και το πρώτο. Ε, είναι παλιό το ζήτημα και είναι και πολύ επικίνδυνο. Το δεύτερο το οποίο ήθελα να αφήξω, το θέμα της εισόδου σε εξυγίανση. Χρειάζεται μεν ευελιξία, για το πότε θα ξεκινήσει αυτή η εξυγίανση. Και είναι σαφές ότι η, ε, η αυτή θα πρέπει να γίνει εγκαίρως. Αυτό που πλευρά μου τι σημαίνει ότι η εξυγίανση θα πρέπει να γίνει πρωτού μα είναι κηρυχθεί αφαιρέγγιος ο κεντρικός αντισυμβαλόμενος, όταν υπάρχουν ακόμα αρκετοί πόροι προκειμένου να γίνει μια τακτική σωστή εξυγίανση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ουσιαστικά συχνά ε, οι κεντρικές συνδεφαλόμενοι έχουν ε, μικρά κεφάλαια και άρα δεν ε, είναι πιθανό να έχουν τεράστιες απώλειες. Η τρίτη κατηγορία έχει να κάνει με τους τρόπους με τους οποίους οι συνομοθέτες θα αποφασίσουν να εναρμονίσουν το πλαίσιο των κεντρικών αντισυμβαλωμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκε ότι οι αντισυμβαλωμένοι είναι πάρα πολύ διασυνδεμένοι και αλληλοεξαρτώμενοι. Η εναρμόνιση λοιπόν με τις ε, η εναρμόνιση της ε, εποπτείας των ε, κεντρικών αντισυμβαλωμένων μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Μία ιδέα θα ήταν προφανώς να επαναλάβουμε την ε, μέθοδο της ε, Τραπεζικής Ένωσης με μια κεντρική, ε, αν θέλετε, αρχή, λαμβάνοντα υπόψη φυσικά ότι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι υπάρχουν σε περιορισμένα κράτη-μέλη, αλλά ειλικρινά οι συλλογικές μας προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν κυρίως προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο της πρότασης πραγματικά οδηγεί σε χρηματοπιστωτική σταθερότητα Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ενδεχομένω να μακρηγόρησα λίγο παραπάνω, Ε, συγγνώμη, και είμαι στη διάθεση σας για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Μέγιορ. Ευχαριστώ, Στίβεν Μαϊτζόρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Ρομπέρτο, που μου έδωσε το λόγο. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Πράγματι, είναι μια θλιβερή ανάμνηση αυτό το οποίο συνέβη πριν ένα χρόνο για τις Βρυξέλλες και την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ για την οργάνωση αυτής της ημερίδας, για τα καθεστώτα ανάκαμψης και εξυγίανσης των κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Θα σας μεταφέρω τις απόψεις μου για τις προτάσεις με βάση τις πρακτικές εμπειρίες της ΕΣΠΑ σε σχέση με την ανθεκτικότητα των CCP όπως γνωρίζετε η σημασία των CCP στην Ευρώπη και παγκόσμια αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια μετά από την εφαρμογή των αποφάσεων του G20 για να αντιμετωπιστούν συστημικοί κίνδυνοι ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Όπως επιβεβαιώθηκε ε, στην άσκηση την οποία οργάνωσε η ΕΣΜΑ πέρυσι, τα CCP συνδέονται με τα μέλη clearing. Γι' αυτό λοιπόν η ε, πτώχευση ενός CCP θα μπορούσε να επηρεάσει σε συστημικό επίπεδο τις αγορές. Η ανθεκτικότητα λοιπόν των CCP είναι βασικό κλειδί για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Τα τελευταία χρόνια η ΕΣΜΑ υποστήριξε την σωστή εφαρμογή της ευρωπαϊκής αντίληψης για την ενίσχυση των αντοχών των κεντρικών αντισυμβαλωμένων έχουμε εμείς ζητήσει να υπάρξει σύγκληση και μέσω κατευθυντηρίων γραμμών και μέσω peer review και μέσω συμμετοχής στα εποπτικά συμβούλια των CCP, τα λεγόμενα Supervisory Colleges. Και έχουμε επίσης οργανώσει stress test για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους και βελτιώνουμε συνεχώς το μεθοδολογικό μας πλαίσιο. Επίσης ελέγχουμε ε, προληπτικά τα CCP όταν αλλάζουν ε, τα πρότυπα κινδύνου για τα ίδια τα CCP. Νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για μια επιτυχή διαδικασία για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τις χρηματαγορές που θα πρέπει να συμπληρωθεί από ένα σαφές πλαίσιο εξυγίανσης που θα διασφαλίσει την βιωσιμότητα των CCP, των κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Γι' αυτό λοιπόν η νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθορίζει ένα ε, πλαίσιο εξυγίανσης των CCP που αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους. Η πρόταση είναι θα έλεγα αναλογική άλλων νομοθετικών ρυθμίσεων όπως της οδηγίας για την εξυγίανση των τραπεζικών ε, ιδρυμάτων, σύμφωνα και με τα ισχύοντα παγκόσμια. Θα ήθελα να εκφράσω λοιπόν την ε, εκτίμησή μου για το, για το ότι οι προτάσεις σας είναι σημαντικές για την ΕΣΜΑ ε, που είναι υπεύθυνη για τις εποπτικές διαδικασίες επί των κεντρικών αντισυμβαλωμένων ίσως να διαφωνήσω με τα συμπεράσματα των προτάσεων ότι όλες αυτές ε, οι επιπλέον αποστολές που μας δίδονται δεν έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις. Είναι σημαντικό να έχουμε τους απαιτούμενους πόρους για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα οποία μας ζητούνται. Καταρχάς τώρα, ε, προγραμματισμός της εξυγίανσης είναι ένα θέμα σημαντικό και θα περάσω στα άλλα ε, μετά. Όταν μιλάμε για τον προγραμματισμό της ανάκαμψης ε, θα υπογραμμίσω τον κεντρικό χαρακτήρα των CCP να κάνουν προτάσεις, ε, προγράμματα εξυγίανσης σύμφωνα με την επίβλεψη των τοπικών ελεγκτικών εποπτικών αρχών όπως επίσης και των Supervisory College. Νομίζω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να βελτιωθεί με πιο ε, συγκεκριμένες τεχνικές λεπτομέρειες έτσι ώστε να υπάρξει εποπτική σύγκληση ε, όπως επίσης και καλύτερη, στο εσωτερικό της Ένωσης όπως και καλύτερη συνεργασία ε, με εξωτερικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπηρεσίες. Δεύτερον, θα ήθελα να δούμε λίγο ε, τα μέσα που προτείνονται στην πρόταση. Είναι βασικό να κατανοήσει κανείς ότι υπάρχουν κάποια παράλληλα σχήματα με τις ε, προτάσεις της οδηγίας για την ανάκαμψη των πιστοτικών ιδρυμάτων, αλλά παρόλα αυτά τα ε, χαρακτηριστικά των CCP είναι διαφορετικά από τα αντίστοιχα των πιστοτικών ιδρυμάτων και των επενδυτικών σχημάτων. Γι' αυτό λοιπόν στο συγκεκριμένο πλαίσιο μην το αγνοήσετε αυτό και πέραν τούτου να υπογραμμίσω ότι τα μέσα τα οποία προτείνονται στην ομοθετική πρόταση επιτρέπουν στις αρχές εξυγίανσης να έχουν το απαιτούμενο επίπεδο ευελιξίας ανάλογα με τις συνθήκες και τη συγκυρία των αγορών. Τρίτον, η διακυβέρνηση της διαδικασίας επίλυσης και εξυγίανσης. Ξέρετε ότι μιλάμε για οργανισμούς και εταιρείες οι οποίες λειτουργούν διασυνοριακά. Ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρχει σωστή συνεργασία ανάμεσα στις εποπτικές αρχές των διαφόρων χωρών. Και εδώ ε, πρέπει να δούμε και ποιος είναι ο ρόλος των λεγόμενων supervisory colleges. Και έχουμε συγκεκριμένες εμπειρίες. Η ΕΣΜΑ μέχρι τώρα δεν τη συζητήθηκε να ξεκινήσει μια διαδικασία διαιτησίας για την μη κατάληξη σε γνωμοδότηση κάποιων τέτοιων supervisory colleges. Για να υπάρξει μια απόφαση από ένα τέτοιο college πρέπει να υπάρχει ε, άνω των δύο τρίτων πλειοψηφία για, το τελικό, για την τελική πρόταση. Αλλιώς προσφεύγουν στην έσμα, κάτι το οποίο όπως είπα δεν έχει συμβεί. Οι υπόλοιπες αρχές στα supervisory colleges όπως τα μέλη clearing πρέπει να προστατεύονται στα πλαίσια της πρότασης την οποία κάνετε. Παρακαλώ αυτό να το λάβετε υπόψη σας όταν διαπραγματεύσετε, διαπραγματεύεστε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέει ότι κάθε μέλος μπορεί να παραπέμπει στην ΕΣΜΑ προς διαιτησία τις προτάσεις επί των οποίων έχει δυσκολία. Νομίζω ότι θα πρέπει να χαμηλώσουμε το επίπεδο δυσκολίας ε, για την κίνηση της διαδικασίας διατησίας. Και τέλος θέλω να μιλήσω εδώ για τη συμβατότητα συγγνώμη, με τα διεθνή επίπεδα. Η πρόταση για την εξυγίανση και ε, ε, ανάκαμψη είναι κάτι που θα πρέπει να είναι συμβατό με τους διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με το ίδιο θέμα. Επιβεβαιώθηκε αυτό στο παρελθόν και πρέπει να επιβεβαιωθεί και στο μέλλον. Να σας διαβεβαιώσω λοιπόν ότι η ΕΣΜΑ κάνει κάθε προσπάθεια για την αποκατάσταση της σταθερότητας χρήματα χρηματαγορές. Νομίζουμε ότι αυτή η σημαντική νομοθετική πρόταση θα πρέπει να πετύχει. Σας ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος και τώρα θα συνεχίσουμε Μάλλον θα αρχίσουμε τη συζήτηση. Και πρώτος ο συνεισηγητής, Ιάκωβος Φον Βάιτσέκερ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσά για τις χρήσιμε παρατηρήσεις. Τρεις ερωτήσεις. Πρώτη. College of Regulators και η προσέγγιση που ακολουθείτε για τους CCP για την ε, ανάκαμψη και εξυγίανση των κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Γενικά τα συστήματα αυτά λειτουργούν πολύ καλά σε καλές εποχές. Βέβαια μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσχέρειες και γι' αυτό άλλωστε φτιάχνουμε και την ε, ε, Τραπεζική Ένωση σε δύσκολες εποχές. Όταν μιλείτε για super majority και άλλα είναι και ένα ζήτημα εμπιστοσύνης όμως που έχει σχέση και με το bond sharing και ποιος πληρώνει ποιο πράγμα εν τέλει. Η πρώτη μου ερώτηση, λοιπόν, λόγω της φύσεως του προβλήματος και ελπίζω ποτέ κανείς από εμά να μην ζήσει ε, την εποχή μιας μαζικής πτώχευσης ενός μεγάλου κεντρικού αντισυραβαλωμένου, παρόλα αυτά θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοια περίπτωση. Και αν συμβεί αυτό, δεν θα υπάρχουν κάποια σειρά επιχειρήματα να ακολουθήσουμε τον δρόμο του ενιαίου επόπτη, single supervisor. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερη, ε, κάπως ευαίσθητη για να το πω και πριν από το τέλος του μηνός, αλλά ας μην το λησμονούμε, έχει σχέση με κάτι που αναφερθήκατε εσείς προηγουμένως, αλλά σιωπηρά, δηλαδή τη Βρετανική έξοδο, το Brexit σε ποιο βαθμό θεωρούμε ότι οι τρέχουσες προτάσεις και αυτές που θα συμπεριληφθούν στον κανονισμό ΕΜΙΡ αλλά και στην πρόταση για ανάκαμψη και εξυγίανση μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ενδεχόμενες προκλήσεις του Brexit όπου ε, δέχεται να έχουμε ε, μίζονες κεντρικούς αντισυμβαλωμένους σε βασικούς τομείς που θα λειτουργούν εκτός της δικής μας δικαιοδοσίας και τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Δεν θα ήταν τουλάχιστον σόφρον να περιληφθεί και ένα στέρεο σύστημα ισοδυναμίας τρίτης χώρας και ενδεχομένως και κάτι σαν αυτό που κάνουν οι Αμερικανοί, δηλαδή να πάμε ακόμα περισσότερο και να επιβάλλουμε κάποιες απαιτήσει εξοδαφικότητας. Τρίτη ερώτηση, πιο συγκεκριμένα για την κυρία Κόνικ τι θα πρέπει να προκαλεί την είσοδο, ξεκινώντας δηλαδή από την αποκατάσταση προς την εξυγίανση, να περάσει δηλαδή σε αυτή τη φάση, γιατί αυτό μπαίνει και σε ένα διαφορετικό πλαίσιο και έχει σχέση και με τις εμπειρίες από το ΕΜΙΡ, δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε τα πράγματα αυτά πριν να φτάσουμε στον καταράκτη waterfall, αλλά θα χρειάζεται ένας αξιόπιστος μηχανισμός που να διασφαλίζει ότι η εξυγίανση δεν, η φάση της δηλαδή δεν αρχίζει υπερβολικά νωρίς. Ότι ο CCP δεν μπαίνει υπερβολικά νωρίς στην φάση της εξυγένσης. Προτιμάτε ερώτηση-απάντηση. Όχι, όλες μαζί. Καλά, τότε να ακούσουμε την κυρία Σουίνμπερν. Μα, εγώ έχω πολλές ερωτήσεις όμως και να με συμπαθάτε. Κυρία Κρένικ, σας ευχαριστώ για την δουλειά που έχετε κάνει για το ψήφισμα FSP δύσκολο ώστε όλοι οι παγκόσμιοι ρυθμιστές να συμφωνήσουν με τα συμπεράσματα. Κάτι σαν αυτό που κάνουμε και εμείς και προσπαθούμε να συμφωνήσουν και πάνω στις ίδιες γραμμές όλα μας τα μέλη. Έχετε την πλήρη κατανόησή μου. Επίσης, αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για μια συνολική πρόταση που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παραμείνει εντός του πλαισίου. Και ω συνεισηγήτρια στόχο μου είναι ότι και εμείς οι πολιτικοί άντρε και γυναίκες να ακούσουμε τους τεχνικούς εμπειρογνώμονε και να μην προσπαθήσουμε να αλλάξουμε πολλές από τις τεχνικές πτυχές της ε, προτάσεως. Αλλά βέβαια έχουμε κάποια μεγαλύτερη διακριτική ευχαίρεια. Τώρα, ερωτήσει για την κυρία Αφού το FSP ε, προσεγγίζει το, την εξυγίανση των, των CCP με ένα είδος εργαλειοθήκης για τα non-default σενάρια είναι διαφορετική η μεταχείριση από τα default σενάρια και εφόσον είναι δεδομένο ένα σενάριο default πάυσης πληρωμών θεωρείται ότι οι δομές κινήτρων επηρεάζονται από ορισμένα από αυτά. Και το άλλο είναι το ζήτημα της Αντισταθμιση ή αποζημίωση. Είμαι βεβαία ότι στο δεύτερο πάνελ θα το συζητήσουμε αυτό, διότι είμαι βεβαία ότι ο κλάδο ε, γνωρίζει ε, πολύ καλά και έχει απόψεις γι' αυτό. Τι μπορείτε να μας πείτε και προς τα πού κατευθύνεται και ιδίω σε ποιο σημείο θα πρέπει να ισχύουν τα μέτρα αποζημίωση. Για τον κύριο Μαϊόρ. Προσέγγιση εργαδιοθήκης για την αποκατάσταση και εξυγένση. Πολύ λίγα περιλαμβάνονται για το δεύτερο επίπεδο της εξυγένσης. Όμως πρέπει να ληφθεί υπόψη και η σημαντική απόκληση μεταξύ των 17 κεντρικών αντισυμβαλωμένων που έχουν έγκριση λειτουργία τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρείτε ότι κάποια σύγκριση είναι δυνατή ή με άλλο τρόπο. Μπορεί να μπουν σε ένα εθνικό σύστημα. Cash equity Ντανούτα Χίπνερ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλες και όλους για τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Συμφωνώ μαζί σας ότι αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι και ένα σημαντικό ελίπον τμήμα του μοσαϊκού στην ε, ρυθμιστική μας αρχιτεκτονική. Και το ίδιο ε, συμβαίνει και πρέπει να προσέχουμε τις διασυνδέσεις ε, και με άλλα τμήματα της νομοθεσίας. Από την άλλη μεριά πρόκειται και για μια ευκαιρία μιας αλλαγής νοοτροπίας ας πούμε. Δηλαδή είναι μια ευκαιρία να προσεγγίσουμε τα πράγματα, ορισμένα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Έχω διάφορες μικρές ερωτήσεις που θα σας υποβάλω. Πρώτα, για την interface μεταξύ του καθεστώτος των τραπεζών και αυτό του CCP. Για, ε, μιλώ πάντοτε για αποκατάσταση και εξυγένση. Από το FSB περιμένουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές πριν αρχίσουμε το σοβαρό έργο επί της εξυγένσης των ε, κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Αλλά πιο ειδική ερώτηση τώρα που έχει σχέση με το γεγονό υπάρχει ένα είδος αρχής του FSB για μη διάκριση CCP τραπεζών που το έχουμε ήδη για την EBRD θεωρείται ότι είναι αρκετό ε, στα πλαίσια μιας παγκόσμιας τραπεζικής κρίσης η οποία θα έχει επιπτώσεις και στους κεντρικούς αντισυμβαλωμένους. Και τώρα η guidance του FSP έχει σχέση και με την διασπορά πληροφοριών μεταξύ CCP και αρχών. Δεν νομίζω ότι στην πρόταση της Κομισιόν υπάρχει τίποτα ειδικά για το θέμα αυτό. Θεωρείτε λοιπόν ότι χρειάζεται κάποια πρόβλεψη για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ CCP και αρχών που είναι αρμόδιες για την εξυγένση, για τον κύριο Μαϊόρ. Θα έχετε δύο επιτροπές εξυγίανσης, μία στην EBA και EBRD Και το άλλο, στο άρθρο 5 του κανονισμού της ΕΣΜΑ. Βλέπετε εκεί κάποια, κάποιο πλεονέκτημα η EBA, ΕΣΜΑ, Επιτροπή να ενταχθεί σε αυτό το σύστημα. Και η δέσμευσή σας που είχα καταλάβει ότι αναλάβατε πριν από ένα χρόνο περίπου και για το haircutting, γιατί πολλοί λίγοι ένας από τους πολύ λίγους, ίσως και ο μοναδικός, ήσασταν πέρσι που είδε το αρχικό περιθώριο του κουρέματος να μην αποκλείεται καταρχήν από την εργαλειοθήκη. Αλλά ορισμένοι το θεωρούν ως ιστάτη καταφυγή, όταν πλέον έχουν ασκηθεί όλες οι άλλες δυνατότητες εξυγένσης. Αυτό δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση της Κομισιόν. Νομίζω όμως το συζητεί το FSB. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, έχει κλείσει πια συζήτηση για το αρχικό περιθώριο του κουρέματος. Εμένετε στην άποψη αυτή και αν ναι, τι είδους ρήτρε διαφύλαξης θεωρείτε ότι μπορούμε να επιβάλλουμε και να χρησιμοποιήσουμε. Ευχαριστώ να μην υπερβαίνει τα τρία λεπτά. Ευχαριστώ και τους κύριους Μάτζο και την κυρία Κένιχ. να αναφερθώ στο, στην εργαλειοθήκη στην οποία ήδη αναφέρθηκε η κυρία Σουίνμπορν και την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ευελιξία από τη μία και την ταχύτητα από την άλλη. Ε, είναι απαραίτητο ένα τέτοιο toolbox, μια τέτοια εργαλειοθήκη, αλλά αν είναι πάρα πολύ δεσμευτική τότε φοβάμαι ότι στο τέλος αν θέλει κάποιος να αντισεβαστεί, όλο και κάτι θα διαφεύγει, όλο και κάτι θα πηγαίνει άσχημα <clears throat> και δεν θα έχουμε το, επιθυμητό αποτέλεσμα, το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να διασφαλίσουμε και την απαιτούμενη ευελιξία έτσι ώστε να διασφαλίζουμε σε ένα δεύτερο επίπεδο την ταχύτητα που απαιτείται γιατί η ανάγκη για ταχύτητα είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση στην περίπτωση της ε, ανάκαμψης, εφόσον μιλάμε για ανάκαμψη. Γιατί αλλιώς υποχρεωτικά θα περάσουμε στην επόμενη φάση ε, της ανάκαμψης. Γι' αυτό λοιπόν και σχετικά με τις παρατηρήσεις Major για την διακυβέρνηση των διαδικασιών ανάκαμψης, ε, πώς θα διασφαλίσουμε την ταχύτητα στη δράση, την ταχύτητα στην αντίδραση, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για μια ουσιαστική αξιολόγηση της κατάστασης ε, με συνέπεια την δυνατότητα λήψης των κατάλληλων μέτρων. Βιέχας. θα ήθελα να κάνω μία θα έλεγα βασικού τύπου παρατήρηση. Βρισκόμαστε στην αρχική φάση. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ξεκάθαρα ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος. Αυτό το οποίο θα ήθελα να ακούσω περισσότερο σχετικά με τους κεντρικούς αντισυμβαλωμένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο συστημικός κίνδυνος τον οποίο εμπεριέχουν και τους οποίους έχουμε ήδη καταγράψει. Θα ήθελα λοιπόν κάποια περισσότερα στοιχεία ε, και για τη συμπεριφορά τους στο πρόσφατο παρελθόν. Ε, έχουν διακινδυνεύσει, ε, αντιπροσωπεύουν ένα συστημικό κίνδυνο ή όχι. Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες λοιπόν γύρω από αυτό. Δεν υπάρχει εδώ θέμα μόχλευσης βέβαια και στην περίπτωση μιας πτώχευσης είναι προφανές ότι θα υπάρξουν ζημίες αλλά η επιμόλυνση η οποία μπορεί να υπάρξει είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει. Ευχαριστώ, δεν υπάρχουν άλλοι. Θα δώσω το λόγο τώρα στη Χέλγα Κόνιγκ. Α, όχι, η έχει ζητήσει το λόγο και αμέσως μετά την ερώτησή σου θα διακόψουμε ε, γιατί όπως είπα θα πρέπει να πάμε στην είσοδο της Ολομέλειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις δύο αυτές παρουσιάσεις οι οποίες ε, μας επέτρεψαν να εξετάσουμε προσεκτικά την πρόταση της Επιτροπής. Τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη ε, τέθηκε ήδη από την Κέιτ Σουίνμπερν Ίσως είναι μια ερώτηση η οποία στρέφεται περισσότερο στον κύριο Μάιτζορ. Μία από τις προκλήσεις που παρουσιάζει η εξέταση της πρότασης της Επιτροπής από το Κοινοβούλιο είναι η μείωση του εύρους, αν θέλετε, ε, δράσης των εθνικών εποπτικών αρχών στην διαδικασία εξυγίανσης. Και αν ναι, ε, ποιοι είναι οι βασικοί οδοί τους οποίους καλούμεθα να εξετάσουμε. Δεύτερη ερώτηση. Έχετε ασκήσει επανειλημμένα κριτική στην λειτουργία των supervisory colleges. Είπατε ότι σε σχέση με την διαδικασία εξυγίανσης ε, τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα για τους κεντρικούς ε, συμβαλόμενους, αντισυμβαλόμενους. Και τέλος πάνω από όλα αυτά τα θέματα και είναι η τρίτη ερώτηση είναι το Brexit. Το ανέφερε ήδη ο Φον Βάιτσεκερ. Πέρα λοιπόν από τις ομιλίες σας, πώς εσείς βλέπετε αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει η Ευρώπη τον 27. Ξέρω ότι δεν είναι η βασική σας αρμοδιότητα, αλλά είστε προσεκτικοί παρατηρητές των κινδύνων για την σταθερότητα των αγορών πώς μπορούν οι εποπτικές αρχές να οργανωθούν σε σχέση με τους συστημικούς κινδύνους τους οποίους ενέχουν οι ε, κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι. Μπορούμε να έχουμε ας πούμε μια διάκριση ανάμεσα στο θέμα του τόπου της αγοράς και στον τόπο καταγραφής ε, της, ε, του συγκεκριμένου αντισυμβαλόμενου, ο οποίος προχωρά σε clearing με ευρώ αποκλειστικά. Σας ευχαριστώ. Τέθηκαν λοιπόν περίπλοκες ερωτήσεις. Θα είναι μια πρόκληση να απαντήσετε σε όλες αυτές, δεν έχετε και πολύ χρόνο. Διακόπτουμε παρακαλώ τώρα, θα επανέλθουμε στις, στις 10 και 5. Πάμε λοιπόν για το ενός λεπτού σιγή μπροστά στην Ολομέλεια. Dear colleagues, please. Λοιπόν, καθίστε συνάδελφοι. Dear Vice Chair, Co-Rapporteur, hello. hello. So, a lot of good questions. Τέθηκαν πολλές και καλές ερωτήσεις. Η κυρία Κιόνικ θα ξεκινήσει τις απαντήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι τέθηκαν πολλές καλές ερωτήσεις. Ίσως ε, ε, για το θέμα του Supervisory College. Να μην ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο συζητάμε εδώ Το θέμα είναι εδώ να εξετάσουμε το σενάριο ε, εξυγίανσης ε, και τι γίνεται με ε, κάποια μέλη clearing και πώς μπορεί το φαινόμενο αυτό να μεταφερθεί σε ευρύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ε, χρειάζεται το college αυτό, διότι θα πρέπει να υπάρχει συνομιλητής και της αρμόδιας αρχής των κρατών μελών για την εξυγίανση και η άποψη των CCP ε, έτσι ώστε ε, ε, να υπάρχει σωστός προγραμματισμός. Σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται μία συζήτηση η οποία δεν θα πρέπει να περιορίζεται αν θέλετε μόνο στα στοιχεία διαφωνίας αλλά θα πρέπει να λειτουργεί και στην δυνατότητα ορισμού ενός αντικειμενικού και μη προκατηλημένου ενδιαμέσου. Είχαμε την πρώτη ε, διαιτησία ε, στην Ευρωπαϊκή Πιστοτική Αρχή. Ε, νομίζω λοιπόν ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτή και μπορείτε να το ελέγξετε. Τώρα εγώ για το Brexit δεν θα πω κάτι συγκεκριμένο σε αυτή τη φάση. Να πω ότι έχουμε διεθνείς CCPs και εντός και εκτός Ευρώπης Οπότε θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι τα CCP στα οποία ανταγωνίζονται το ένα το άλλο ε, ανταγωνίζονται στο ίδιο επίπεδο ασφάλειας έκθεσης σε κίνδυνο και ότι θα πρέπει να υπάρχει διασταυρούμενη αναγνώριση των καθεστώτων μέσα στα οποία λειτουργούν έτσι ώστε να μην τίθενται θέματα ασυμβατότητας και νομίζω ότι το να υπάρχουν ισχυροί CCP σε συγκεκριμένους τομείς είναι κάτι το θετικό. Τώρα, τι μπορεί να προκαλέσει την είσοδο στη διαδικασία εξυγίανσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε πει επανειλημμένα. Σαν αρχή επί της εξυγίανσης απαιτείται ευελιξία. Ταυτόχρονα έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο δείχνει ότι τη στιγμή που ξεκινά στη διαδικασία εξυγίανσης ε, στην ουσία εισέρχεσαι ε, σε ε, περιουσιακά δικαιώματα θα έλεγα διαφορετικών μερών, διαφορετικών και πολλών εμπλεκομένων. Οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις και χειρότερες καταστάσεις από ό,τι ας πούμε στις αντίστοιχες περιπτώσεις για τις τράπεζες. Στην ουσία λοιπόν ε, αυτό το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ε, απολύτως δεσμευτικά αλλά είναι κατευθυντήριες γραμμές. Αν ένας κεντρικός αντισυμβαλόμενος δεν είναι σε θέση να αποκαταστήσει ε, την βιωσιμότητά του, τότε θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι διαδικασίες θα ακολουθήσουν. Και εδώ ε, τίθενται σε συζήτηση τα θέματα των μέσων αποκατάστασης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κεντρική αντισυμβαλόμενη δεν είναι πιστοτικά ιδρύματα. Είναι στην ουσία ένας μεγάλος υπολογιστής ο οποίος θα πρέπει να λειτουργεί συνέχεια έτσι ώστε να προχωρά στα απαιτούμενα clearing και γι' αυτό απαιτούνται ε, κάποια μέσα ανάλογα με το πρόβλημα το οποίο τίθεται οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις ε, για την εξυγίανση είναι οι προσπάθειες αποκατάστασης της βιωσιμότητας των εταιριών αυτών, αποκατάστασης των θέσεων τις οποίες κατέχουν, όπως επίσης τίθενται στην επόμενη φάση και το θέμα της κατανομής των ζημιών ανάμεσα στα μέλη του clearing και ακόμα και ευρύτερα. Αυτό που απαιτείται λοιπόν για μία αρχή επί της εξυγίανσης είναι να έχει τη διάθεσή της ε, τα μέσα τα οποία προβλέπονται για την ανάκαμψη των CCP έτσι ώστε να παίρνει άμεσα αποφάσεις. Οι αποφάσεις θα πρέπει ε, να λαμβάνονται όσο είναι ακόμα καιρός. Τώρα το θέμα των αποζημιώσεων. Το FSP δεν έχει ακόμα πάρει αποφάσεις. Σκόπιμα θα έλεγα. Ε, δεν έχει εφαρμόσει τις προτάσεις που εφαρμόζονται σε επίπεδο τραπεζικών ιδρυμάτων. Υπάρχει πάντα σύνδεση ανάμεσα στο CCP και στα μέλη clearing που θα πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις που πρέπει. Στην περίπτωση όμως που κατανείμει στις ζημίες είναι σαφές ότι θα πρέπει να εκχωρηθούν κάποια ε, δικαιώματα ιδιοκτητικά Εδώ δεν θέλω να ασκήσω κριτική στα μέτρα τα οποία προτείνουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην εργαλειοθήκη. Απαιτείται όμως ευελιξία και δυνατότητα αν θέλετε μέτρων που θα αποκαταστήσουν την ισορροπία. Και για μια άλλη ερώτηση, αν έχουμε να κάνουμε με συστημικούς κινδύνους. Έχουμε αποδείξεις από το παρελθόν γι' αυτό όχι, δεν έχουμε τέτοιες άμεσες αποδείξεις. Αλλά παρόλα αυτά, ε, τα όργανα αυτά καθίστανται προοδευτικά όλο και πιο συστημικά. Οπότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τι θα συμβεί αν μία από τις ε, μεγάλες αυτές εταιρείες ε, αποτύχει, πτωχεύσει. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό, να μην το ζήσουμε αυτό, αλλά παρόλα αυτά δεν έχω να πω κάτι άλλο στην παρούσα φάση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις αυτές που κάνατε αξιότιμοι βουλευτέ της επιτροπή ΕΚΟΝ και να απαντήσω. Καταρχάς, υπάρχουν πολλές ερωτήσεις για το θέμα της ευελιξίας και της αναλογικότητας αφενός και της ταχύτητας. Και τι γίνεται σε ό,τι αφορά την πρόταση εξυγίανσης. Ε, θεωρώ ότι το σημαντικό είναι να αντιληφθούμε ότι αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι ευελιξία και αναλογικότητα μεν, αλλά σε ό,τι αφορά τα παράγωγα και την εξυγίανση είναι ένα θέμα το οποίο υπόκειται σε μεγάλο ανταγωνισμό και θα υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα και θα, και θα υπάρχουν και άλλοι παραγοντέ. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ναι μεν υπάρχει αναλογικότητα και ταχύτητα, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτό ως μια πρόκληση για, για μεσολάβηση και διατησία μεταξύ επιχειρήσεων. Και γι' αυτό λοιπόν είπαμε και είπα και εισαγωγικά ότι θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη καθοδήγηση για τα εργαλεία εξυγίανση και ανάκαμψη, γιατί θεωρούμε ότι αυτό θα βοηθούσε σε ό,τι αφορά την συνοχή και την ομοιογένεια. Και αυτό είναι ο λόγο που είπαμε ότι θα πρέπει να μειώσουμε καθώς τον πύχη σε ό,τι αφορά την, ε, την αίτηση και την εκκίνηση της διατησίας και διαμεσολάβησης και η εμπειρία μας μας ε, καταδεικνύει αυτό ακριβώς. Σε τρία χρόνια δεν έχουμε ούτε μία περίπτωση ουσιαστικά τέτοια ε, διαιτησία. Είναι σημαντικό λοιπόν και είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι το γεγονό ότι κάτι παραπέμπεται στην ΕΣΜΑ δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα πάρει ε, πολύ χρόνο η λήψη απόφασης. Στο παρελθόν έχουμε δει και αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί σε 24 ώρες. Ε, είναι τεχνική η αντιμετώπιση και ξέρουν ότι θα πρέπει να δώσουν λοιπόν γρήγορα μια απάντηση. Να αποφύγουμε λοιπόν τον ανταγωνισμό μεταξύ των ε, ρυθμιστικών συστημάτων και να περιορίσουμε και τα εμπόδια για την αναπομπή στην ΕΣΜΑ. Κατά πόσον τώρα θα πρέπει να περάσουμε σε μια ενιαία εποπτεία και κατά πόσον ε, υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος να είναι αρκετά ισχυρός και στεναρός. Αυτό που θα ήθελα να διευκρινίσω στο σημείο αυτό, μιλώντας ως τεχνοκράτης, τα τεχνοκρατικά επιχείρηματα τα οποία προβάλλονται για την κεντρική εποπτεία είναι αρκετά στεναρά και πιστικά θα ήταν πιο ισχυρό ο μηχανισμό αν ήταν ενιαία η εποπτεία. Εκ παραλλήλου, φυσικά με τη μέθοδο που έχουμε τώρα με τα διάφορα σώματα, το σύστημά μα είναι πιο ισχυρό από ό,τι ήταν πριν το ΕΜΗΡ. Άρα, κοιτάξτε, είναι πολιτική η απόφαση, δεν είναι τόσο τεχνοκρατική, γιατί τα τεχνικά επιχειρήματα για μια κεντρική εποπτεία είναι μάλλον συντριπτικά. Τρία επιχειρήματα θα ήθελα να αναφέρω στο πλαίσιο αυτό, κοιτώντα και τα σχετικά επιχειρήματα για μια κεντρική επιχειρήση ε, εποπτεία, συγγνώμη. Καταρχάς, η αλληλοσυνδεσιμότητα. Συνδεσιμότητα. Όχι μόνο με του κεντρικού συνδεσιμαλόμενους, αλλά και με το τραπεζικό σύστημα. Ύστερα, όπω σα είπα, υπάρχει μεγάλος πειρασμό ε, ανταγωνισμού για την κανιστικό πλαίσιο. Και τρίτον, σε ό,τι αφορά την οικονομία των προσόντων. Να αντιληφθούμε ότι μετά τον Brexit θα υπάρχουν 13 CCPs ε, ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί εξ αυτών θα είναι υπό την εποπτεία μια αρχής και μόνο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μεγάλη ικανότητα εποπτείας και είχαμε ήδη μια περίπτωση όπου η αρχή αυτή εποπτείας ανέθεσε την εποπτεία στην ΕΣΜΑ. Τώρα, η συζήτηση που συνεχίζεται για τις τρίτες χώρες και τις πολιτικές τους στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο υπό τον υφιστάμενο μηχανισμό ισοτιμίας υπάρχουν δυνατότητε εποπτείας οντοτήτων σε τρίτες χώρες. αλλά είναι υπερβισμένε δυνατότητε να συζητηθούν, για παράδειγμα, από του CCP τρίτων χωρών και να εφαρμοστούν και αποφάσει. Αυτό φυσικά αποτελεί μια πολύ περιορισμένη δυνατότητα. Και το έχουμε αναλύσει αυτό και στο παρελθόν. Θα είναι σημαντικό να σκεφτούμε κατά πόσο χρειαζόμαστε πιο καλούς μηχανισμούς και σε τι βαθμό εξασφαλιζόμαστε ότι ο νομοθέτης της τρίτης χώρας λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους που δημιουργεί ενδεχομένως ο CCP της χώρας στην Ευρωπαϊκή ε, περιοχή, επικράτεια. Προς το παρόν δεν υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια ευθύνη επισήμω για να ληφθούν ε, υπόψη οι κοινωνικοί κανόνες. Τώρα, για τις δύο διαφορετικές επιτροπές ε, εξυγίανσης στην EBA και στην ΕΣΜΑ. Αυτό που προσπαθήσαμε να τονίσουμε και εισαγωγικά, εγώ τουλάχιστον, είναι το εξή. Η εξυγίανση των CCP διαφέρει εκ από την εξυγίανση των τραπεζών. Είναι διαφορετικέ οι δομέ ιδιοκτησία, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά θέματα πληροφόρηση και τι θέσει. Είναι πολύ διαφορετικά πράγματα. Ξέρετε ότι στι τράπεζε, για παράδειγμα, είναι δύσκολο να έχει κανεί αξιόπιστε πληροφορίε και για... όλα αυτά είναι πολύ λιγότερο προβληματικά, αν θέλετε. Είναι πιο απλά σε ό,τι αφορά τα CCP. Άρα θεωρώ ότι υπάρχει λόγο να υπάρχουν δύο επιτροπέ. Από την άλλη, υπάρχουν και αρκετέ ε, δικλείδε ασφαλείε ε, στην προτάση προκειμένου να υπάρχει σωστή ανταλλαγή απόψεων μεταξύ EBA και ΕΣΜΑ. Τώρα, για τα πρεθόρια διαφοροποίησης και τα κουρέματα κτλ. Α, προβλέπεται η δυνατότητα κουρέματος ε, αρχικών περιθωρίων μάλλον ε, περιθωρίων διαφοροποίηση, όχι αρχικών περιθωρίων όμως. Θέλουμε να έχουμε εργαλεία στην εργαλειοθήκη μας. Καταλαβαίνουμε φυσικά όμως και το επιχείρημα ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ομοιογένεια και στο διεθνές επίπεδο. Καταλαβαίνουμε την απόφαση που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο αυτό για να μην εντοπιστούν ρήτα τέτοιοι μηχανισμοί. Τέλος, για τους συστημικούς κινδύνους των CCP. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε πόσο ότι χρειάζεται να λειτουργούν μάλλον ήδη λειτουργούν υπό αυστηρούς όρους και χρειάζονται σωστά περιθώρια ε, και ανταποκρίνονται στους κανόνες δύο μέλων εξυγίανσης, το οποίο είναι ήδη μια σημαντική υποχρέωση. Είναι ανθεκτική λοιπόν η CCP. Παράλληλα, αυτέ οι δοκιμέ αντοχή, τα stress test, δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Είναι σε φάση επεξεργασία ακόμα και κοιτάμε τον κίνδυνο αποτυχία των ομολόγων. Θα κοιτάξουμε και του κινδύνου στα επόμενα τεστ τη ρευστότητα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και πρόεδρο. Και τώρα να περάσουμε στο δεύτερο πάνελ τη ακρόαση μα. Ε, θα δώσω την Προεδρία στην Κέι Σουίμπορν. Σας ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη στο σημείο αυτό προς τον πρώτο αντιπρόεδρο που κάθεται δίπλα μου. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την ακρόαση αυτή. Για το χρονοδιάγραμμα να σας πω δύο λόγια. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη προβλέπεται στις 11 και ως μία από τις συνεισηγητρίες θα μιλήσω λίγο λιγότερο. Αν θα μπορούσατε να περιοριστείτε στα 5 έω 6 λεπτά, ε, αν θα μπορούσατε να περιοριστείτε λίγο λοιπόν, για να έχουμε λίγο πιο πολύ χρόνο και για τις ερωταπαντήσεις. Και επίσης να ζητήσω από του κοιόδης και από τον συνεισηγητή να έχουμε 2 λεπτά για ερωτήσεις και μετά να δώσουμε τον ε, λόγο στους Πανελίστε πάλι για να απαντήσουν και να τελειώσουμε πριν από τι 11. Για να μην καθυστερούμε λοιπόν, θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Ερικ Μιούλερ CEO της Eurex Clearing, να πάρει το λόγο. Ο πρώτος ομιλητής από πλευρά του κλάδου, του οικονομικού κλάδου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμοι βουλευτές, αξιότιμοι, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Οίκων. Να ευχαριστήσω και την ε, Πρόεδρο και τον κύριο Βαϊτσέκερ που διοργάνωσαν την ακρόαση αυτή. Μεγάλη τιμή για μένα και για την Eurex Clearing, την ε, εταιρεία την οποία εκπρόσωπο που μας καλείται να συζητήσουμε σήμερα μαζί σε αυτό το σημαντικό θέμα. Προτού περάσω στην ευρωπαϊκή πρόταση την κάθε αυτή, να κάνουμε λίγα βήματα προς τα πίσω, να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή και να υπενθυμίσουμε γιατί συζητάμε σήμερα το φάκελο αυτό. Πριν από 10 χρόνια η μεγαλύτερη οικονομική κρίση από το 1929 ξεκίνησε και παρά το γεγονός ότι όλοι έχουμε κουραστεί ε, να το λέμε και να το ακούμε, θεωρώ ότι πρέπει να το επαναλάβουμε, ότι η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 έθεσε σε κίνηση τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση, το μεγαλύτερο οικονομικό τέλμα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η παροχή τέτοιων ε, μεθόδων και μέσων αρρωγής ανταποκρίνεται στο 100% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Και έτσι λοιπόν προαπαιτήθηκαν, μάλλον απαιτήθηκε η λήψη έκτακτων μέτρων και αυτό συμφωνήθηκε στο G6 το 2009 στο Pittsburgh. Ωστόσο, αυτές οι αποφάσεις κακώς ε, θεωρούνται καμιάς φορές ε, απλά μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, γιατί υπήρχε και ένας απότερος στόχος. Ο απότερος στόχος λοιπόν ήταν να αποφευχθούν μερικές οικονομικές κρίσεις τέτοιου επίπεδου και να προληφθεί, αν θέλετε, και η ζημιά στο πρωτοφόλι του φορολογούμενου, παρά το γεγονός ότι όλοι είχαμε υπόψη τα όσα συνέβησαν με τα κεφάλαια των τραπεζών. Μία άλλη μεγάλη θρησική απόφαση ήταν να κοιτάξουμε τι γίνεται και με τα OTC derivatives, με τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα. Η οικονομική κρίση λοιπόν αποκάλυψε σε τι βαθμό η έλλειψη διαφάνειας και πληροφορήσεις για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους ε, είχε οδηγήσει σε ένα περίπλοκο και αδιαφανές ε, δίκτυο το οποίο δυσκόλαβε πάρα πολύ τους ε, συμμετέχοντες φορείς να εντοπίσουν το σωστό επίπεδο κινδύνου και έτσι αυτό απειλούσε την οικονομική σταθερότητα. Προκειμένου λοιπόν να βελτιωθεί η αποδοτικότητα, η ακεραιότητα, η διαφάνεια στην αγορά παραγόγων, αποφασίστηκε να ε, εισαχθούν δύο προαπαιτήσεις, δύο ζητήματα. Καταρχάς, να υπάρχει πιο διαφανής τρόπος ε, ανταλλαγή πληροφοριών και κατά δεύτερον υποχρέωση εξυγίανση μέσων κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Όπω ξέρετε, σκοπό τη εξυγίανση είναι αντί ο καθένας ε, να βρά με μυστικό τρόπο κάποιοι φορείς οι οποίοι θεωρούνται ανεξάρτητοι να αποτελέσουν τα σημεία αναφοράς για τις ε, συναλλαγές αυτές και αυτό θα βελτιώνει την διαφάνεια και τη διαχείριση του κινδυνού αφραγγιότητας αλλά επιτρέποντας και την ε, δικτύωση των απολειών αυτών για να κρατήσει το σύστημα από μόνο το πιο αποδοτικό και, παρά και επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θα ήθελα να θέσω τρία σημεία και να αναφερθώ και σε κάποια ζητήματα τα οποία ανέφεραν οι προλαλήσαντε. Καταρχά, το πρώτο που θα πρέπει να γίνει για να υπάρχει μια σωστή δομή παροχής κινήτρων και να αποτραπεί η χρήση των χρημάτων του φορολογουμένου στο μέλλον. Μπορεί να είναι απλό και να φαίνεται απλό, αλλά είναι να εξαιρεθεί η χρήση δημόσιων χρημάτων από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως έχει το κείμενο, περιλαμβάνει στην παρούσα φάση τη δυνατότητα δημοσίας διάσωσης, ε, δημοσίου bailout και αν ε, οι συμμετέχοντες μπορούν να κληθούν να αποζημιώσουν ε, σε ποσοστό μεγαλύτερο της συμμετοχής της, ενδεχομένως να μην υποστηρίξουν την ανάκαμψη και να προτιμήσουν την εξυγίανση στην οποία θα συμμετέχει το κράτος. Και αυτό προφανώς δημιουργεί σε μεγαλύτερο κίνδυνο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ανάκαμψης και εξυγίανσης. Κατά δεύτερον, και με την λογική, θα ήθελα να υπογραμμίσω τους κινδύνους συμπερίληψης ρήτρα αποζημίωσης ε, στην νομοθετική πρόταση. Γιατί αν ένα μέλος εξυγίανσης αξιολογεί την υπηρεσία εξυγίανσης, το όφελο συνέχισης αυτής. Γιατί να αποζημιώνεται λοιπόν το μέλος αυτό α, για τη συμμετοχή του. Αν αποζημιωθεί η απώλεια ενός συμμετεχόντος φορέα, ο οποίος έχει συμφωνήσει σε θελούσιο επίπεδο για την κατανομή απώλειών προκειμένου να παρέχονται βασικές υπηρεσίες, η συνέπεια είναι η κατανομή χωρίς απώλειες ενδεχομένως κάποιοι να θεωρήσουν, μάλλον πιστεύουμε τα ωφέλη της ε, συνέχισης της παροχής αυτών των κρίσιμων υπηρεσιών είναι ήδη πάρα πολλά και ενδιαφυσβήτητα και πέρα από τα προφανή ωφέλη. Αυτή η συνέχιση παροχής υπηρεσιών επιτρέπει και στους συμμετέχοντες να συνεχίσουν να βγάζουν έσοδα από την παροχή υπηρεσιών εξυγίανσης από τους πελάτες, να μειώσουν τις ε, γραφές για το κεφάλαιο και να υπάρχει και κόστος αντικατάστασης ενδεχομένω. Αυτά είναι μόνο κάποια παραδείγματα των ωφελών. Κάτι άλλο που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Από πού θα προέλθουν τα χρήματα αν ε, τα ίδια κεφάλαια των CCP αν δεν αρκούν αυτά τα χρήματα η απάντηση φυσικά είναι προφανή. Ο φορολογούμενο. Και αυτό με οδηγεί στο τελευταίο σημείο. Την αρχή του ότι δεν θα πρέπει να επιδεινώνεται η θέση των μισθωτών σε σχέση με την αφαιρεγκαιότητα. Δεν θα πρέπει να είναι περιόριστη αυτή η συμμετοχή, γιατί η αρχή αυτή τι σημαίνει ότι οι αρχές εξυγίανσης θα πρέπει σε τελική ανάλυση με υπεύθυνο τρόπο να βοηθούν. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι θα τους δέσουν ε, χειροπόδαρα τις αρχές αυτές εξυγίανσης σε ό,τι αφορά για παράδειγμα ενδεχόμενο κίνδυνο καταγγελίας αν αποφασίσουν να παρεκκλίνουν από τις κανόνες των κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Άρα θέλουμε έναν ευρύ ορισμό τη αρχή αυτή μη επιδείνωση στη θέση των πιστωτών σε σχέση με την αφαιρεγκαιότητα. Δηλαδή, όταν ένα πιστωτή μετά την εξυγίαση βρεθεί όντω σε χειροτερή θέση, αν έχει ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία αφαιρεγκαιότητα, αυτή η μείωση τη αξία θα πρέπει να αναφέρεται σε όλα, σε όλε τι συνιστώσει ε, της εξυγίανσης σε ό,τι αφορά την απώδεια απώλεια εισόδηματων, την πρόσβαση στα έσοδα, συστημικά ζητήματα. Συνοψίζοντας, ε, μας χαροποιεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρούμε ότι είναι σχεδόν ε, άψογη για την δημιουργία ενός θωρακισμένου συστήματος. Ε, ενισχύει την ανθεκτικότητα και τη διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών μας αγορών, ωστόσο να μην ξεχνάμε γιατί μας έχει διδάξει η τελευταία κρίση. Η πρόταση λοιπόν θα πρέπει να μην περιλαμβάνει καταρχάς τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται δημόσια χρήματα, κατά δεύτερον η δυνατότητα των μελών εξυγίανσης να ζητούν αποζημίωση και τρίτον να καταγγέλλονται ε, οι άρχες εξυγίανσης. Σας ευχαριστούμε και πάλι και για την ευκαιρία αυτή και για τον χρόνο σας και προσβλέπω στη συζήτηση και στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Θα παρακαλέσω τον κύριο Μακκόρμικ που είναι Chief Risk Officer στην τράπεζα BNP. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας να απευθύνω τον λόγο στην Επιτροπή σας για θέματα CCP. Μας ικανοποιεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πριν να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, θα ήθελα να σας αναφέρω ποια πράγματα έχουν ήδη επιτευχθεί. Παρα, θα παρακαλούσουν οι διερμηνείς στον ομιλητή, αν είναι δυνατόν να ακούει κάποιος να του πει να μιλάει λίγο πιο αργά, διαβάζει πολύ γρήγορα. Βεβαίω, εξυγίανση τη τράπεζα δεν σημαίνει πτώχευση, ότι δεν συνεπάγεται πτώχευση. Εδώ χρειάζεται αναλογικότητα και βεβαίω αυτή είναι αποτελεσματικότερη. Περισσότερα πράγματα μπορούν να γίνουν για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις αυτές. Οι τράπεζες πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούν ξανά και ξανά. Δηλαδή, Πέρα από την αναλαγωγικότητα νομίζω ότι η πρόταση η οποία γίνεται πρέπει να διασφαλίζει την διαφάνεια έτσι ώστε να είναι επιτυχής ε, και να είναι πράγματι η ανάκαμψη μια ουσιαστική και σταθερή διαδικασία. Ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να ορίσει συγκεκριμένους αντικειμενικούς δείκτες και η είσοδος στην διαδικασία εξυγίανσης δεν θα πρέπει να θεωρείται κάτι το, κατά το αναπόφευκτο. Σχετικά με τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους, αυτοί θα επιλέγουν τη στιγμή κατά την οποία θα πρέπει να εισέλθει κάποιος στην ανάκαμψη, στη διαδικασία ανάκαμψης. Τα μέλη clearing θα πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς από ποια στιγμή και μετά εκτίθενται στις κρίσεις οι οποίες τους περιβάλλουν. Θα πρέπει να ελαττωθούν τα επίπεδα αβεβαιότητα στο ελάχιστο δυνατό. Προς λοιπόν της διαφάνειας θα πρέπει να υπάρχουν ε, συγκεκριμένες διαδικασίες και για τα προγράμματα ανάκαμψης όπως και τα προγράμματα εξυγίανσης. Θα πρέπει όλα αυτά να λαμβάνονται υπόψη λοιπόν από τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία της διαχείρισης κινδύνου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Καταρχάς το επίπεδο της τρέχουσας έκθεσης. Δεύτερον, ε, θα πρέπει να είναι γνωστό το ανώτατο επίπεδο ζημιών που μπορεί να προκληθούν, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν οι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι. δεν θα πρέπει οι ζημίες ε, να ξεπερνούν τα όρια τα οποία έχουν καθοριστεί και σε επίπεδο και στην περίπτωση πτώχευσης και στην περίπτωση συνέχισης της δραστηριότητας. Το τρίτη, η τρίτη βασική αρχή είναι η αποτελεσματικότητα. Εμείς θέλουμε να υπάρξει μια απλοποιημένη διαδικασία για μια ανάκαμψη την οποία θα καθοδηγεί ο κεντρικός αντισυμβαλόμενος αυτό θα επιτρέψει την ευελιξία που απαιτείται για την αντιμετώπιση κινδύνων διαφορετικών προφίλ. Η αποτελεσματική ανάκαμψη θα πρέπει να διατηρήσει την αξία των CCP, να διατηρήσει την χρηματοπιστωτική ισορροπία και να ελαχιστοποιήσει τις ζημίες κατανέμοντάς τες με έναν δίκαιο τρόπο θα πρέπει να γίνει σεβαστός ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο αυτός ο οποίος αντιμετωπίζει το πρόβλημα ε, θα πρέπει να κατανέμει τις ζημίες τις οποίες προκαλεί και να μην δημιουργείται επίπεδο επιπλέον ηθικού κινδύνου. Τίθεται το θέμα επίσης και ε, των ε, εργαλειοθηκών. και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται η διαδικασία για να καλύπτονται ζημίες οι οποίες έχουν προκληθεί σε διαφορετικά επίπεδα. Δεν θα πρέπει επίσης ε, να ζητείτε από τα CCP να συμπληρώνουν κενά τα οποία δεν είχαν προβληθεί εκ των προτέρων. Το λεγόμενο initial margin, το αρχικό περιθώριο, είναι αυτό το οποίο θα καθορίζει το πεδίο δράσης ε, των ε, CCPs. Η διαδικασία η οποία λοιπόν ακολουθείται δεν είναι μια επιπλέον διαδικασία παροχής ρευστότητας και θα πρέπει να αντισταθμίζεται η ε, λειτουργία σαν παράδειγμα η εφαρμογή ενός haircut θα πρέπει να αποζημιώνεται η εφαρμογή ενός haircut. Τέλος θα πρέπει οι αμοιβιοποιημένοι πόροι για τα CCP που διατίθενται στην αντιμετώπιση της έκθεσης σε κίνδυνο να μην χρησιμοποιούνται για την ανακεφαλαιοποίησή τους γιατί αυτό θα δημιουργήσει στρεβλά κίνητρα. Ε, προς την κατεύθυνση αυτή η αποζημίωση με τη μορφή μετοχών, ομολόγων μάλλον, των CCP δεν είναι κάτι το κατάλληλο. Να ζητήσω από την κυρία Κίλη και οι τελικοί επενδυτές είναι αυτοί που μας ενδιαφέρουν. Η Άιλιν Κίλι είναι στην BlackRock υπεύθυνη για θέματα αξιολόγησης κινδύνων. Να μου επιτρέψετε να κάνω κάποια σχόλια εμείς προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά τα επενδυτικά σχήματα τα οποία χρησιμοποιούν ας πούμε οι συνταξιούχοι και οι μεμονωμένοι επενδυτές στην Ευρώπη. Προσπαθούμε να δούμε ακριβώς τις συνέπειες που μπορεί να υπάρχουν από διάφορους εξωγενείς παράγοντες. Η BlackRock ε, δεν αναλαμβάνει ίδια τον κίνδυνο απέναντι στους κεντρικούς αντισυμβαλωμένους, οι πελάτες μας τον αναλαμβάνουν. Αλλά εμείς προσπαθούμε να εκπροσωπήσουμε σωστά τα συμφέροντα των επενδυτών και αποταμιευτών. Προσπαθούμε να μειώσουμε τον συστημικό κίνδυνο. Εγώ είμαι επαγγελματίας στον τομέα της διαχείρισης κινδύνου Είμαι μέλος της ομάδας αξιολόγησης κινδύνου αντισυμβαλωμένων της BlackRock. Η δουλειά μου γίνεται σε επίπεδο χρηματοπιστωτικό, προσπαθώ δηλαδή να εντοπίσω και να μετριάσω τους κινδύνους σε επίπεδο πιστωτικό για τους πελάτες της BlackRock. Εμείς σήμερα μιλάμε για ανάκαμψη και εξυγίανση θα πρέπει να σας ζητήσω να μην ξεχάσετε ε, την σημασία μιας άλλης λέξης, της ανθεκτικότητας. Νομίζω ότι θα πρέπει ε, ο κεντρικός αντισυμβαλόμενος να βοηθήσει τους επενδυτές του να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους αν υπάρξουν ε, προβλήματα στις αγορές. Στόχος μας λοιπόν είναι να ενισχύσουμε και την ανθεκτικότητα ενός κεντρικού αντισυμβαλόμενου έχουν αρχίσει να γίνονται οι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι συστημικά σημαντικοί και θα πρέπει να υπόκεινται σε συγκεκριμένες κεφαλαιοχικές απαιτήσεις. Ε, μέχρι τώρα ε, δεν έχει επιμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό. Καταρχάς θα πρέπει το κεφάλαιο των CCP να χρησιμοποιείται για δύο λόγους. Πρώτον, να είναι σε θέση να απορροφήσει α, ζημίες επιχειρηματικές οι οποίες δεν προέρχονται από περιπτώσεις πτώχευσης. Και δεύτερον, σε σχέση με περιπτώσεις πτώχευσης, να χρησιμοποιηθεί σαν μηχανισμός απορρόφησης των ζημιών και να μπορέσει να διαχειριστεί με σωστό τρόπο τις επόμενες φάσεις. Πολλές φορές τα κεφάλαια τα οποία έχουν στη διάθεσή τους ε, τα CCPs θεωρούνται για πολλούς πάρα πολύ λίγα, ενώ οι ίδιοι οι ε, αντισυμβαλόμενοι θεωρούν ότι είναι επαρκέστατα. Ποιο είναι το καλύτερο επίπεδο κεφαλαίων που πρέπει να υπάρχει ε, και τι τίθεται θέμα ηθικού κινδύνου σε σχέση με τους συμμετέχοντες. Πώς θα προσμετρηθεί ο κίνδυνος αυτός. Νομίζω ότι η διασφάλιση της ανθεκτικότητας των CCP απαιτεί ένα υγιές αναλυτικό πλαίσιο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για τους CCP έτσι ώστε η ακρίβεια των πληροφοριών να είναι δεδομένη. Τα CCP που είχαν πολλές φορές μονοπόλιο σε ορισμένες αγορές έχουν θα έλεγα γίνει λιγότερο συστημικά σημαντικοί σε πάρα πολλούς τομείς ε, και πολλές φορές ε, έχουν, ε, υπάρχουν απαιτήσει για δημοσιοποίηση στοιχείων λειτουργίας οι οποίες είναι χαμηλότερες και από κάποιες μικρές εισηγμένες επιχειρήσεις. Τώρα για τα θέματα εξυγίασης και ανάκαμψης. θα πρέπει οι αρχές να είναι σε θέση να ελέγχουν τις διαδικασίες αυτές. Δεν θα ήμουν σήμερα εδώ αν πιστεύαμε ότι οι διαδικασίες είναι πλήρεις. Πιστεύουμε ότι μπορούν να ενισχυθούν έτσι ώστε να προστατευτούν τα συμφέροντα των επενδυτών συνταξιοδοτικών ταμείων και μετά. Θα πρέπει να γίνει η διαφοροποίηση ανάμεσα στους χρήστες, τους τελικούς των διαδικασιών clearing και τους διαχειριστές χρήστες. Η διάκριση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική σε σχέση με τα μέσα τα οποία ε, είναι διαθέσιμα σε έναν κεντρικό αντισυμβαλόμενο. Σχετικά με την ανάκαμψη των CCP πιστεύουμε ότι είναι λάθος να επιτρέψουμε ένα κεντρικό αντισυμβαλόμενο που είναι μια κερδοσκοπική επιχείρηση να παίρνει τα χρήματα του πελάτη αν αποτύχει να παρέχει ακριβώς την μετρίαση του κινδύνου που του ζητήθηκε. Παίρνει τα χρήματα που ανήκουν στους συμμετέχοντες στις αγορές, ε, στους συνταξιούχους, από τους συνταξιούχους και τα χρησιμοποιεί για να καλύψει τις ζημίες που είναι καρπός ε, της αποτυχημένης διαχειριστικής ε, διαδικασίας. Αυτό είναι κάτι που μας ανασυχεί λοιπόν. Καταρχάς, μιλάμε για τρεις σημαντικές έννοιες. Έλεγχος. Ο έλεγχος έρχεται στην περίπτωση κατά την οποία οι πόροι οι διαθέσιμοι έχουν εξαντληθεί. Οπότε μόνο οι αρμόδιες αρχές για την ανάκαμψη και την εξυγίανση θα είναι σε θέση να κατανείμουν τις ζημίες δεν θα πρέπει οι ίδιοι οι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι αλλά οι αρμόδιες αρχές να ελέγχουν τις επιπτώσεις της δράσης του συγκεκριμένου αντισυμβαλωμένου στην πραγματική οικονομία. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των ελεγκτικών αρχών να ξεκινήσουν την διαδικασία κατανομής των ζημιών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει συγκεκριμένη αρμοδιότητα των ελεγκτικών αρχών. Τα ανώτατα όρια τώρα, αν οι αρμόδιες αρχές θεωρούν ότι το haircutting θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν μέσο κατανομής ζημιών, θα πρέπει αυτό να γίνεται για να προστατευθούν τα οικονομικά συμφέροντα του συστήματος και των τελικών επενδυτών μπορεί να επιβληθούν σαν παράδειγμα ανώτατα όρια και ποσοτικά για το ίδιο το haircut ή και για την χρονική διάρκεια του haircut. Και η τρίτη βασική έννοια είναι η αποζημίωση. Όλοι οι τελικοί χρήστες από την ανάκαμψη ή την εξυγίανση ενός τελικού αντισυμβαλόμενου θα πρέπει να αποζημιωθούν πλήρως από τον ίδιο τον αντισυμβαλόμενο. Οι τελικοί επενδυτές θα πρέπει να τύχουν προτεραιότητας πιστοτικής σε σχέση με τα ποσά που χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης. Το καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι το, αρχι, το, το αρχικού περιθωρίου δεν θα πρέπει να επιτρέπεται και για την ανάκαμψη και για την εξυγίανση, γιατί συνεισφέρει στο εύθραυστο του συστήματος. Σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας και σας υπενθυμίζω ότι έχουν υποβληθεί και γραπτά ε, σχόλια και θα υποβληθούν στην διαπραγματευτική ομάδα. Θα ήθελα να αρχίσω τώρα λέγοντας αν θέλει ο συνεισηγητής Ιάκωβ Φων Βάιτσέκερ να θέσει ερωτήσεις. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και θα περιοριστώ έτσι σε μόνο μια ερώτηση και στις ε, τρεις τοποθετήσεις σας δείξατε την ε, μεγάλη περιπλοκότητα των ε, contingent liabilities, των ευθυνών που προκύπτουν από την πρόταση που έχουμε μπροστά μας. Βεβαίως και αυτό είναι τμήμα της δουλειάς σας, αυτό είναι απόλυτα κατανοητό. Ο κάθε προσπαθεί να τοποθετηθεί ε, με έναν τρόπο ώστε να βελτιώσει κάπως ε, την θέση του μέσα σε αυτήν την ε, ρύθμιση για τις ευθύνες. Αυτό που με ανησυχεί εμένα είναι ότι αν πάρει κανείς την περιπλοκότητα αυτή συν την περιπλοκότητα του benchmark ότι δηλαδή κανένας πιστοτίζει θα πρέπει τελικά να βρεθεί σε ε, επιδεινωμένη θέση. Είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ όποιος δηλαδή επιτύχει κάποια ε, περιθωριακά κέρδη. Αν μιλούμε για ένα πραγματικό σενάριο αρμαγεδόνος, όπου μπαίνουν σε πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση ε, παραπάνω από ένας CM, θα έχουμε και στο επίπεδο του οργανισμού που εμπλέκεται, αλλά και στο πολιτικό επίπεδο, να προωθήσουμε αυτή την πάρα πολύ περίπλοκη ρύθμιση για contingent liabilities και τελικά θα επιβάλλουμε ένα τεράστιο βάρος στους φορολογουμένους. Ερώτηση, δεν θα ήταν πολύ ευκολότερο, πολύ απλούστερο να έχουμε υψηλή ικανότητα απορρόφησης ε, ζημιών, για παράδειγμα υψηλό ποσοστό κεφαλαίου σε CCP, επίσης υψηλό κεφάλαιο σε CM, όπου όλοι αυτοί οι παίκτες και παγκόσμια να έχουν υψηλή κεφαλαιοποίηση για να μπορούν να αποζημιώνουν τους πελάτες, κάτι το οποίο θα μειώσει και σημαντικά, δραματικά την περιπλοκότητα του συστήματος. Δεν θα έπρεπε λοιπόν στόχος μας να είναι η προσπάθεια περιορισμού του, ε, της περιπλοκότητας για να ε, μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτό το σενάριο Αρμαγεδόνος που ε, αναφέραμε πριν. Ε, η κυρία Σουίνμπουρν, θα θέσω κι εγώ μια ερώτηση για το περιθώριο για το κούρεμα, που για μένα είναι από τα πιο αμφισβητούμενα σημεία και αυτό που με κάνει εμένα να δυσκολεύομαι περισσότερο. Ήμουν και εισηγητής έκθεση ιδία πρωτοβουλία του 2013 εδώ στο Κοινοβουλίο, που είχαμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το εργαλείο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό την αιγίδα της ε, αρχής εξυγίανσης. Έχουμε τώρα ρύθμιση που περιλαμβάνει την δυνατότητα χρήσης αυτού του εργαλείου μέσα στα πλαίσια της εξυγίανσης, επομένως μέσα στα πλαίσια του rulebook των CCP και όχι μόνο υπό την έγκριση της ε, αρχής εξυγίανσης. Σημαντική αλλαγή. Πρέπει να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί και γιατί έχει φτάσει και υπέφτασε. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη ή τις απόψεις των ε, πανελίστ πώς προβλέπετε την χρήση του ε, haircut ε, στο σύνολο των κανόνων, στο rulebook που εφαρμόζεται και πώς χρησιμοποιείτε. Το χρησιμοποιείτε με τον ίδιο τρόπο όπως και άλλοι CCP. Για τον κύριο από την PNB Paribas. Θα χρησιμοποιήσει το ίδιο με το VMGH για τους πελάτες σας και για τα CCP εκείνα που χρησιμοποιούν στα rulebook τους το VMGH. Σας έχουν εξηγήσει την προσέγγιση που επιλέγουν και εξηγείτε στους πελάτες σας τι σημαίνει για αυτούς όπως είναι σήμερα. Και τέλος για την BlackRock, τους τελικούς χρήστες. Ποιες προφυλάξεις βάζετε για την χρήση του VMGH για την εξηγένση. Ευχαριστώ. Επανέρχομαι τώρα στην κυρία Χίπνερ που θα υποβάλει ερώτηση. Θα κάνω κάτι που δεν θα έπρεπε ποτέ να κάνω, δηλαδή θα θέσω την ερώτηση μου και αναγκαστικά θα αποχωρήσω μετά. Αλλά θα παραμείνει βεβαίω η συνεργάτη μου για να ακούσει την απάντηση. Δύο ερωτήσει μάλιστα. Μία αναφέρεται στο βασικό στοιχείο του, της, ε, ε, αποκατάστασης και εξυγίανσης για τα περιουσιακά στοιχεία. Η ρύθμιση που έχουμε είναι παρόμοια με αυτήν που έχουμε στην BRRD, εξωτερική δηλαδή αξιολόγηση. Αλλά υπάρχουν και μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε τράπεζες και CCP σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση. Αν πάρετε για παράδειγμα στην EBRD για τα παράγωγα έχουμε πληροφορίες για τα παράγωγα που παρέχονται από τους CCP, για παράγωγα δηλαδή τα οποία συμψηφίζονται. Αυτό όμως δεν συμβαίνει εδώ για την εξήγηση των CCP. Οποιοδήποτε σχόλιο από εσά θα το εκτιμήσω. Πώς βλέπετε δηλαδή την αξιολόγηση, πώς μπορεί να διεξαχθεί. Δεύτερη ερώτηση για, το, για τα όσα είπε ο κ. Μίλλερ Πρόκειται πράγματι για απολύτω στεγανή πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμω στο χρηματοπιστωτικό τομέα πρέπει να αναζητούμε και λύσει οι οποίε ε, να είναι στεγανέ και για του μελλοντικού κινδύνου. Και ε, για τον ε, κλάδο εδώ, ο οποίο αναπτύσσεται, σχεδιάζουμε έναν κανονισμό που αντιμετωπίζει το τρέχον πλαίσιο και το παρελθόν, αλλά γνωρίζετε πολύ καλά ότι ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές σε ό,τι αφορά νέα περιουσιακά στοιχεία που θα χρειαστούν νέους μηχανισμούς και να αντιμετωπιστούν και οι ρυθμίσεις που γίνονται μεταξύ πελατών και μελών του συστήματος. Άρα εκεί θα χρειαστεί κάποια ευκαμψία για το μέλλον. Ερώτηση. Βλέπετε αυτή την ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη ευκαμψίας που όλοι κατανοούμε, αλλά και ασφαλείας δικαίου από την άλλη μεριά με την πρόταση φτάνουμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο στην ισορροπία αυτή ή χρειάζεται βελτίωση της ισορροπίας κατά την άποψή σας. Σας ευχαριστώ πολύ για το ανοιχτό πνεύμα με το οποίο ε, απαντήσατε ως τώρα. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε και πίεση χρόνου. Η κόρα που είναι και η τελευταία ε, σκιώδη συγγήτρια. Μάλιστα αισθάνομαι και εγώ την πίεση. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω τους άλλους πανελίστ να αντιδράσουν για το τμήμα εκείνο της ε, ανθεκτικότητας ε, για το θέμα που έθεσε η BlackRock. Γιατί από εκεί ξεκινούν όλα. Ίσως μπορούν και οι άλλοι να απαντήσουν σε αυτό. Υπάρχει ήδη κάποια ανάλυση, υπάρχει ε, κάποιο ιστορικό, κάποιες πληροφορίες, κάποιο background. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλες και συζητητές. Ας επιστρέψω το μικρόφωνο λοιπόν στα μέλη του πάνελ. Αν θέλετε να Επιλέξτε κάποια ερώτηση για να απαντήσετε. Σας παρακαλώ σε δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που δίνετε την ευκαιρία να απαντήσουμε σε ορισμένες από αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Θα ήθελα να αρχίσω με την ερώτηση για το κεφάλαιο η οποία ακούστηκε μια-δυο φορές. Είναι πολύ σημαντικό όταν εξετάζει κανείς του CCP να αντιλαμβάνεται πού βρίσκονται οι γραμμές άμυνας. Και το πιο σωστό είναι η κατάλληλη, η κατάλληλη αξιολόγηση της διαχείρισης του κινδύνου που πρέπει να έχει μια δομή. Θεωρούμε ότι είναι σωστό το νομοθέτημα. Είναι διαφορετικό από αυτά που κάνουν οι τράπεζες και νομίζουμε επίσης ότι είναι και πιο εξειδικευμένο από ό,τι θα δείτε σε οποιοδήποτε άλλο θύλακο ε, συμμετεχόντων, είτε asset manager τραπεζών είτε και σε άλλους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Το EMIR εξετάζει ακριβώς αυτό. Ένας μεγάλος ECP όπως η Eurex θα έχει περιθώριο περίπου 50 δισεκατομμυρίων το περιθώριο λοιπόν επιτρέπει τη διαχείριση του κινδύνου και είναι ο βασικός παράγοντας που επιτρέπει την απορρόφηση των ε, κραδασμών στο σύστημα. Και η στάθμιση του περιθωρίου για να μπορεί να αντιμετωπίζει τους κραδασμούς αυτούς, όπως για παράδειγμα, μπορεί να είναι πολύ σημαντική, όπως η κρίση της τράπεζας Λέμαν και τα όσα μπορεί να συμβούν με το Brexit. Είναι σταθμισμένο λοιπόν το περιθώριο ώστε να μπορεί να αντέξει τους κραδασμούς. Equity capital, το ε, μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί ε, να παίξει τον ρόλο αυτού του εργαλείου διαχείρισης κινδύνου. Το άλλο σημαντικό εργαλείο είναι ίσπραξη και πληρωμή variation margin. Οι μηχανισμοί αυτοί αποτελούν και τον πυρήνα τη καθημερινή μα δραστηριότητα από την πλευρά του κεφαλίου. Πρέπει να είναι κανεί πολύ προσεκτικό σε ό,τι αφορά τα κίνητρα που δίνει. Όσο περισσότερο μετοχικό κεφάλαιο απαιτείται να καταθέτουν οι CCP, λιγότερη συμμετοχή θα νιώθουν οι συμμέτοχοι, διότι η απορρόφηση κρατασμών να λαμβάνεται από κάποιον άλλο. Για να μην διακινδυνεύσει λοιπόν αυτή η δομή των κινήτρων είναι σημαντικό να βρεθεί μια ισορροπία και θεωρούμε ότι ο κανονισμός ΕΜΗΡ έχει βρει αυτή την ισορροπία. Και για την Eurex Clearing εμείς μπορώ να πω ότι έχουμε ευχαριστώς ε, υιοθετήσει όλες τις απαιτήσεις και μάλιστα και παραπάνω από ότι ε, με συγχωρείτε πολύ θα αναγκαστώ να σας διακόψω γιατί πρέπει να δώσω δύο λεπτά και στους υπολείπους από δύο λεπτά. Και ο επόμενος ομιλητή μας περιμένει έξω από την αίθουσα. Για το GNGS βλέπουμε ότι το εργαλείο εξυγίανσης θα έπρεπε να να είναι στα χέρια της αρχής εξυγίανσης. Και αυτό θα είναι υπό την ηγεσία των CCP. Μας ρωτήσατε επίσης κατά πόσον θα διαβιβαστεί ο κίνδυνος στους πελάτες, αν χρειαστεί. Νομίζω ότι αν φτάσουμε στο σημείο αυτό, νομίζουμε ότι όλοι οι παράγοντες της χρηματοπιστωτικής αγοράς θα πρέπει να συμμετέχουν, να συμμετέχουν στην εξυγένση. Άρα ναι, για την πιο απλοποιημένη προσέγγιση τώρα των CCP, των επιπέδων κεφαλαίου των CCP. Νομίζω ότι αυτά τα δύο συνδέονται. Θα πρέπει να αποφύγουμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση χρήσης όλων των πόρων που έχουν χρησιμοποιηθεί αν υπάρχει λοιπόν σωστή διαφάνεια, θεωρώ ότι αυτό από μόνο το πατάει ένα τμήμα της ερώτησης. Η κυρία Κέλλη, συγγνώμη. Να προσπαθήσω να απαντήσω στις δύο ερωτήσεις. Καταρχά, στο VGMEH. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την εξυγίανση, ποτέ ε, για ανάκαμψη των ε, κεντρικών αντισυμβαλωμένων κατά πόσο μας έχουν ε, ενημερώσει το DHM, Image είναι τμήμα του της εργαλειοθήκης. Εγώ και η ομάδα μου κοιτάξαμε τους κανόνες ε, των CCP για να το βρούμε και εμείς οι ίδιοι, δεν ξέραμε. Και γι' αυτό λοιπόν ε, αυτό είναι το αντικείμενό μου, αλλά δεν είναι και απλό να σας πω την αλήθεια. Κατά δεύτερον, το θέμα της πόλης σύνθετότητας στην οποία αναφέρατε. Διδάσκω θέματα εξυγίανσης σε πολύ κόσμο. Και ένα πράγμα που λέω συνέχεια είναι ότι είναι πάρα πολύ πολύ σύνθετο το θέμα αυτό. Γιατί πλέον η ομολογία για δεν είναι δύο, είναι πέντε. Θα ήθελα λοιπόν να απλοποιηθεί κάπως η κατάσταση. Αυτό θα πρέπει να το πετύχουμε. Δυστυχώς όμως μας προκαλεί πονοκέφαλο σε όλους μας, μην νομίζετε. Ευχαριστώ. Θα ήθελες να μιλήσεις, ε, Γιάκοπ, ένα-δύο λεπτά για να συνοψίσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε χρόνο στους συναδέλφους που θα το κοιτάξουν το θέμα αυτό. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν που ήλθατε εδώ και μας βοηθήσατε πάρα πολύ πραγματικά. Και νομίζω ότι διευκρινίστηκαν οι τομείς στους οποίους θα πρέπει να δώσουμε προσοχή εμείς ως συνομοθέτες. Κάποια θέματα είναι θεσμικά, που έχουν να κάνουν με τη διασυνοριακή φύση των δραστηριοτήτων. Ένα άλλο ζήτημα έχει να κάνει με την περιπλοκότητα. Ναι, δεν μπορούμε να την αποφύγουμε, αλλά θα πρέπει παρόλα αυτά να κατανοήσουμε ε, καλύτερα αυτά που κάνουμε και τι είδου κίνητρα δίνουμε εξάντε σε ό,τι αφορά την κατανομή των απολύων στους CCP, στους φορολογούμενους, στους πελάτες και στις τράπεζες και ίσως θα έπρεπε να τα λέμε και λίγο πιο ξεκάθαρα αυτά, χωρίς να περιορίσουμε φυσικά υπέρ του την ευελιξία όπου αυτή χρειάζεται, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε κάπως πόσο εφαρμόσιμε θα ήταν αυτές οι λειτουργίες σε μια πραγματική κρίση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάκο. Ευχαριστώ. Σαν συνεισηγήτρια και πρόεδρος έχω την τελευταία λέξη, δεν μου συμβαίνει συχνά. Έχει σημασία να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια που έχει γίνει από τότε που ξεκινήσαμε με την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Νομίζω ότι η προσπάθεια που κάναμε ήταν πρωτοποριακή και είναι πλέον μια προσπάθεια αναφοράς και είστε πλέον οι εμπειρογνώμονες και σε σχέση με τις υποδομές των αγορών και σε σχέση με την προληπτική αντιμετώπιση των χρηματαγορών. Ε, γι' αυτό λοιπόν η βελτίωση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν είναι κάτι το αναμενόμενο και νομίζω ότι σαν πολιτικός εγώ δεν μπορώ να προτείνω φυσικά ε, τις τεχνικές ρυθμίσεις, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε το ποιος είναι αυτός ο οποίος εποπτεύει τις χρήσεις των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν. Να πω επίσης ότι η διαπραγματευτική ομάδα ε, παρέχει κίνητρα για όλους τους συμμετέχοντες ε, και ενώ τους αντισυμβαλωμένους και γι' αυτό το ΕΜΙΡ νομίζω είναι ένα πολύ καλό πλαίσιο και στην ουσία αυτό που κάνουμε τώρα είναι να συνεχίσουμε αυτά τα οποία προβλέπονται στο ΕΜΗΡ και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκλίνουμε από τους κεντρικούς άξονες των αποφάσεών μας στο παρελθόν. Έχει μεγάλη σημασία για μας να κατανοήσουμε ότι η σωστή και συνεχιζόμενη διακυβέρνηση σε εισαγωγικά των κεντρικών αντισυμβαλωμένων είναι θα έλεγα αυτό το οποίο θα διασφαλίσει και την ανθεκτικότητά τους. Θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να δούμε ε, κατά πόσον η ανταπόκρισή μας είναι αναλογική. Οι διάφορες, ε, ε, υπάρχουν διάφοροι τύποι κεντρικών αντισυμβαλωμένων στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Κάποιες είναι μικρές και εξειδικευμένες, κάποιες είναι γενικότερης χρήσεως και ευρύτερες. Γι' αυτό η νομοθετική αυτή πρόβλεψη θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με αναλογικό τρόπο, έτσι ώστε να μην βασίζεται σε ονομαστική, αν θέλετε, διάκριση, αλλά σε σχέση με το επίπεδο του κινδύνου. Και τώρα, πού είναι η γραμμή, πού είναι το σύνορο ανάμεσα στην ανάκαμψη και την εξυγίανση. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να καθοριστεί με αποφασιστικό τρόπο ή αν απαιτείται να υπάρχει μια ενδογενής ευελιξία στο σύστημα το οποίο να είναι σε θέση να διακρίνει και να επιλέξει το ένα πεδίο ή το άλλο. Κλείνοντας ως ο πρόεδρος και ως συνεισηγήτρια λέγοντας ότι έχουμε πάρα πολλές τεχνικές ομάδες οι οποίες θα συνεδριάσουν γύρω από το θέμα αυτό και η διαπραγματευτική ομάδα θα μπορέσει να κατανοήσει καλύτερα το τι επιθυμούν οι εμπλεκόμενοι και να μπορέσουμε να δούμε από πού προέρχονται οι ανησυχίες και ποιες είναι οι πιθανές λύσεις. Θα ήθελα να ενθαρρύνω λοιπόν όσους ε, θέλουν να πάρουν μέρος στη διαδικασία αυτή να ενημερωθούν για τα χρονοδιαγράμματα. Θα υπάρχουν και στην ιστοσελίδα της ΕΚΟΝ και γι' αυτό αν θέλετε να μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας. Δεν θέλουμε να αποκλείσουμε κανένα και θέλουμε η διαπραγματευτική μας ομάδα να είναι όσο πιο ευρύτερη γίνεται ε, και να εκπροσωπεί όλους τους εμπλεκομένους και τις ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές ε, και τις ε, κρατικές υπηρεσίες. Το συγγνώμη από το πάνελ για τον χρόνο τον περιορισμένο Έχουμε τα γραπτά σας σχόλια, θα ανταλάβουμε υπόψη σας και να είστε σε επαφή με την διαπραγματευτική ομάδα διμερός εάν θέλετε να τονίσετε κάποια συγκεκριμένα επιμέρους σημεία. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Νομίζω ότι πλησιάσουμε στην τελική φάση έτσι ώστε ε, να βελτιώσουμε την ανθεκτικότητα των κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Just to inform members who are here, we have Mr. Να σας ενημερώσω ότι έχουμε τον κύριο Κωνικοπής που με τον πρόεδρο, τον κύριο Κουαλτιέρη. Θα έρθουν σε λίγο.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 Dear ε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, απευθύνω το καλό ορίσατε στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων, κύριο Χόιερ, Τον ευχαριστώ για την παρουσία του εδώ, για ακρόαση για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Έχουμε παράδοση πλέον ανταλλαγής απόψεων μεταξύ της Οικονομικής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που θα εορτάσει τα 60 της χρόνια το 2018 και που ε, είναι ανεξάρτητης ό,τι αφορά την λήψη αποφάσεων μέσα στο σύστημα αλλά και έχει και το στρατηγικό ρόλο για την χρηματοδότηση επενδύσεων στις χώρες μέλη. Ε, στα πλαίσια αυτά το προσωπικό της και ο πρόεδρός της συμμετέχουν σε συζητήσεις με τις ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει εκθέσεις ελέγχου των δραστηριοτήτων της τράπεζας και των λογαριασμών της. Διεξάγουμε την ε, συζήτηση αυτή με τον κύριο Γόιερ σε πολύ επίκαιρη στιγμή, διότι πρόκειται να ψηφίσουμε την έκθεση για τις δραστηριότητε της ε, Τράπεζας Επενδύσεων με εισηγητή τον κύριο Κίρτσο. Θα γίνει αυτό το, στη σημερινή απογευματινή συνεδρία και έχουμε αρχίσει ήδη τις συζητήσεις και για το νομοθετικό φάκελο για το ΕΦΣΙ και έχει υποβληθεί και έκθεση από την Δευτέρα. Αγαπητέ Πρόεδρε, καλώς ήρθατε και σας δίνω τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, με χαρά επιστρέφω μπροστά σας. Όταν κάποιος είναι εκτός κοινοβουλίου, σαν μέλος ε, για πέντε χρόνια, πρέπει να προσπαθήσει να ανακάμψει σε επίπεδο κοινοβουλευτικού DNA. Γιορτάζουμε τα 60 χρόνια και θα υπάρξει και η συγκεκριμένη συνάντηση στη Ρώμη το Σαββατοκύριακο. Τον επόμενο χρόνο θα γιορτάσουμε τα 60 χρόνια της τράπεζας είναι μια ανεξάρτητη δομή στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οργάνων. Είναι αληθές βέβαια αυτό κατά κάποιο τρόπο, αλλά τα κράτη-μέλη μας ελέγχουν σε σχέση ανεξαρτησίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της οποίας τη σύμφωνη γνώμη χρειαζόμαστε για κάθε πρόγραμμα μικρό και μεγάλο, μας ελέγχει και αυτή. Και εσείς είστε ο βασικός μας συνομιλητής όταν προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε μια χρηματοδοτική βάση σε σχέση με αυτά τα οποία κάνουμε και σε σχέση με την απελευθέρωση των κεφαλαίων Θα μιλήσουμε και για το ΕΦΣΙ σήμερα. Σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε πετύχει πολλά σήμερα. Υπάρχουν θετικά και αρνητικά σε σχέση με τις εξελίξεις αλλά υπάρχουν και τρόποι για την περαιτέρω βελτίωση των μέσων τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Χωρίς όμως την θαραλέα απόφαση των συνομοθετών και αυτών που είναι υπεύθυνοι για τα θέματα του προϋπολογισμού να θυσιάσουν 16 δις σε σχέση με άλλα προγράμματα όπως το Horizon 2020 δεν θα μπορούσαμε να ελέγξουμε το ΕΦΣΥ το οποίο είναι πραγματικά και νέο αν θέλετε μέσο σε σχέση με τους ε, πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας, τα δάνεια και τις εγγυήσεις που μπορούμε να διαθέσουμε. Είναι λοιπόν ένα υπαδειγματικό νομίζω βήμα σε επίπεδο δημοσιονομικό, σε επίπεδο βελτίωσης των δαπανών και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά υπάρχει όμως και χώρος ε, βελτίωσης. ο λόγος ύπαρξης αν θέλετε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι η στήριξη της συνοχής και η ε, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς μέσα από ε, επενδυτικά μέσα, μέσα από επενδυτικούς τρόπους ενισχύουμε την ανάπτυξη και δημιουργούμε ε, θέσεις απασχόλησης εκεί όπου υπάρχει ανεπάρκεια. Συνεπώς λοιπόν στην ουσία λειτουργούμε συνολικά. Πριν, συζητήσω, πριν έρθω στην αίθουσα εδώ, αναφερθήκαμε ότι θα πρέπει να πάρουμε κάποιες οδυνηρές αποφάσεις ε, για το Ηνωμένο Βασίλειο, σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Μιλάμε για 22 δις ε, ε, τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν αποθεματικά στην τράπεζα γιατί εμείς δεν κατανέμουμε φυσικά τα κέρδη και ε, τα σορεύουμε στους ιδίους πόρους τους οποίους έχουμε στη διάθεσή μας. Τα κράτη-μέλη λοιπόν έχουν πληρώσει μόνο 22 δις. Αν προσέξετε ε, θα έχουν, έχουν εισπράξει 12 δις. Γιατί ε, όπως σας είπα τα αποθεματικά μετατρέπονται σε κεφάλαιο. Συνεπώς λοιπόν με 12 δις ευρώ τα οποία έχουν εισπράξει τα κράτη-μέλη με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα βιβλίο δανειοδότησης που έχει φτάσει τα 600 δις περίπου. Ε, πραγματικά το πλεονέκτημα αυτό αυξάνεται για τα κράτη-μέλη και την επιχειρηματικό κόσμο σε ετήσια βάση είναι κάτι το οποίο ξεπερνά τις κεφαλαιοχικές ενέσεις οι οποίες μπορεί να έχουν γίνει προς κάποια κράτη-μέλη. Είναι ένα πολύ ισχυρό μέσο, πρέπει λοιπόν να το εξηγήσουμε καλύτερα, πρέπει να το δημοσιοποιήσουμε καλύτερα γιατί το μέγεθος ε, της δραστηριότητάς μας είναι διπλάσιο από την Παγκόσμια Τράπεζα. Έχουν τα κράτη-μέλη δηλαδή ε, μέσα πραγματικά ουσιαστικά για την καταπολέμηση των κρίσεων. Και γι' αυτό λοιπόν η τράπεζα μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες της. Θυμηθείτε ότι όταν ο πρόεδρος Γιούνκερ προσπαθούσε να να θα έλεγα γλύψει τις πληγές του μετά από τις τελευταίες εκλογές στο Λουξεμβούργο ε, είχε τεθεί το ερώτημα τι θα κάνω αν με εμπιστευθούν να είμαι ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Εμείς αναλύσεις κάναμε στην τράπεζα. Έχουμε ένα πολύ ισχυρό οικονομικό τμήμα προβλέψεων και του είπαμε να δει τα τους περιορισμούς σε επενδυτικό επίπεδο στην Ευρώπη. Βέβαια τα επιχειρήματα εδώ έρχονται από τη μία και από την άλλη σε σχέση με τους αντικειμενικούς αριθμούς. Αλλά παρόλα αυτά μπορεί κανεί να δει τους στόχους τους οποίους θέτει το Συμβούλιο και να συγκρίνει τους στόχους αυτούς με τις πιστώσεις οι οποίες προβλέπονται σε επίπεδο εθνικών και κοινοτικού προϋπολογισμού. Και αυτό εκείνη την εποχή μας οδηγούσε σε μια διαφοροποίηση 700 ε, σχεδόν ε, δις. Για να μην μακρηγορώ τώρα και να πω ότι στα πλαίσια του πρώτου χρόνου λειτουργίας του ΕΦΣΥ έχουμε πετύχει πολλά. Μειώσαμε ε, τα 700 σε 600. φυσικά πετύχαμε κάτι, αλλά είναι ένα τμήμα μόνο της προσπάθειας που πρέπει να γίνει. Πέραν τούτου, αυτή τη στιγμή συζητήσαμε το πρόγραμμα Juncker για πρώτη φορά οι πολιτικοί ηγέτες και στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή πήραν αποφάσεις να υποστηρίξουμε τους στόχους αηφορίας των Ηνωμένων Εθνών, με τους οποίους είχαμε συμφωνήσει. Μερικούς μήνες μετά ε, συμφώνησαν οι πολιτικοί μας ηγέτες και για τους στόχους COP21. Αυτό σημαίνει ότι διευρύνεται αυτό το, ε, το επενδυτικό κενό. Γιατί οι στόχοι τους οποίους θέτουμε και στα πλαίσια του ΚΟΠ και σε σχέση, σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία απαιτούν περαιτέρω επενδύσεις. Γι' αυτό λοιπόν ε, είχαμε πάρει την απόφαση με τη δική σας υποστήριξη τότε και ήταν μια έγκαιρη, εγκαίρος ληφθήσα απόφαση. Να ξεκινήσω λοιπόν βλέποντας ε, ποιο είναι το επενδυτικό περιβάλλον και οι επενδυτικές τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς εμείς ε, και η ομάδα μας βελτιώνει το κλίμα το επενδυτικό στα κράτη-μέλη. Για την εξωτερική διάσταση δεν θα αναφερθώ τώρα, για να μην μακρηγορήσω, αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις αργότερα. Ανακάμπτει λοιπόν η επένδυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η ανάκαμψη δεν είναι ε, η ίδια σε όλες τις χώρες και στις κατηγορίες. Σε κάποιες κεντρικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ε, στο επίπεδο ε, που ήταν πριν από την κρίση. Ενώ σε άλλες χώρες, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, είναι 8% χαμηλότερο από ό,τι ήταν πριν από την κρίση. Υπάρχουν διαφορές στις επιδόσεις. Η ανάκαμψη αυτή δεν είναι μόνο αργή, αλλά είναι πιο αργή από άλλου είδους κρίσεις στο παρελθόν. Βλέπουμε λοιπόν μια κάποια ανάκαμψη, αλλά φαίνεται ότι απαιτεί περισσότερο χρόνο από ό,τι έγινε μετά από άλλες κρίσεις στο παρελθόν. Υπάρχουν περιορισμοί που το δικαιολογούν αυτό. Έχουν μειωθεί οι επενδύσεις σε υποδομές, οι ιδιωτικέ επενδύσεις και αυτές βελτιώνονται αν και είναι χαμηλότερα από τα επίπεδα στα οποία ήταν πριν από την κρίση. Ε, σε κάποιες χώρες ισχυρές ε, έχουν φτάσει τα επίπεδα προκρίσεως, αλλά όχι σε όλες. Γι' αυτό λοιπόν η κατάσταση, αν συγκρίνει κανείς ιστορικά τα στοιχεία, ε, βλέπει ότι δεν είναι ικανοποιητική για την καινοτομία, την δημιουργία θέσεων εργασίας και τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε να κάνουμε με ένα διαφθρωτικό επενδυτικό κενό, στο οποίο αναφέρθηκα και στην εισαγωγή μου. Ε, υπολογίζεται ότι χρειαζόμαστε 100 δις για να βελτιώσουμε τα δίκτυα ενέργειας για την διασφάλιση της παροχής ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές, 80 δις ε, για τις ε, συγκοινωνίες και μεταφορές, 65 δις για να πετύχουμε την ψηφιακή λεγόμενη ατζέντα, όχι μόνο σε σχέση με το ευρύ φάσμα, κάτι το οποίο συζητάμε, αλλά και με το θέμα της αποθήκευσης δεδομένων και την κυβερνοασφάλεια. 10 <coughs> δις ε, για την εκπαίδευση, συν τα 90 τα οποία έχουμε εξοδέψει στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, 90 δις για τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες, τη διασφάλιση παροχής καθαροίδατος και 130 δις για την έρευνα και την ανάπτυξη για να πετύχουμε τον στόχο του 3% του ΓΑΕΠ. Και τέλος, αν δει κανείς ε, την ε, επενδυτική κουλτούρα των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ευρώπη σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε, θα πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις σε επίπεδο venture capital ε, πάνω από 35 δις. Όλα αυτά λοιπόν προστίθενται. Και έτσι λοιπόν, το πόσο επιμένουν τα χάσματα αυτά ε, μας κάνουν να αναρωτιόμαστε για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Και μετά από 10 χρόνια ομφυλοσκόπησης θεωρούμε ότι έχει έρθει πλέον η στιγμή να κοιτάξουμε την Ευρώπη από πλευρά παγκόσμιας οικονομίας και τότε διαπιστώνουμε πόσο γρήγορα κινούνται κάποιοι από τους εταίρους μας. Και έτσι κάναμε μία έρευνα επενδύσεων μεταξύ 12.000 ε, εταιριών, μικρές και μεσαίες για να καταλάβουμε το πώς επενδύουν, τις ανάγκες τους, τις συνήθειές τους. Και η έρευνα λοιπόν επιβεβαιώνει ότι η ανάκαμψη των επενδύσεων είναι, ενισχύεται. Και υπάρχει τάση ενίσχυσης και όχι τόσο ύφεση. Ωστόσο, υπάρχουν και πράγματα που με ανησυχούν. 15% των εταιριών αναφέρουν ότι οι επενδυτικέ του δραστηριότητε τα τελευταία τρία χρόνια ήταν υπερβολικά χαμηλέ για να εξασφαλίσουν την επιτυχία της ε, επιχείρησής τους και την πραγματική ανάπτυξή τους και κατά μέσο όρο ε, λιγότερο από τις μισές θεωρούν ότι ο εξοπλισμός τους είναι σύγχρονος και μόνο 40% θεωρούν ότι ε, πληρούν τις υψηλές προδιαγραφές για την ενέργεια. Σε ό,τι αφορά τις καινοτομίες, οι πιο πολλές επιχειρήσεις προσαρμόζονται στις καινοτομίες, δεν τις προωθούν. Επίσης, σε ό,τι αφορά σε τα εμπόδια για τις επενδύσεις. 69% ε, των επιχειρήσεων εκτιμά ότι αυτός ο γενικός όρος είναι εμπόδιο για τις επενδύσεις τους και επίσης η έλλειψη πεπειραμένου και καταρτισμένου εργατικού δυναμικού αποτελεί ένα συνήθις πρόβλημα στις επενδύσεις. Έχουμε δημογραφικά ζητήματα, θέματα εξωτερικής μετανάστευσης, δηλαδή ανθρώπων που φεύγουν από τις χώρες και αυτό αποτελεί πρόβλημα. Επίσης, ο κανονισμός για, τα, για τις επιχειρήσεις και η νομοθεσία αποτελούν προβλήματα σε διάφορες περιπτώσεις. Η πρόσβαση στην χρηματοδότηση, βασικό θέμα για τις μικρές επιχειρήσεις και κυρίως όταν ε, είναι άειλο το αντικείμενό τους σε ό,τι αφορά και το κόστος χρηματοδότησης και τις απαιτήσει που αντιμετωπίζουν ε, οι επιχειρήσεις αυτές. Ε, το κόστος της χρηματοδότησης ε, είναι πιο υψηλό σε κράτη-μέλη που έχουν πληχθεί από την οικονομική κρίση. Το 75% τη είπα στις επένδυσεις και τη χρηματοδότηση πρόκειται από τι θετικέ αγορέ. Ε, έχουμε μεγάλη διαφορά εδώ πέρα και θα πρέπει να το γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα. Σα είπα λοιπόν τι κάναμε λίγο πολύ. Το 2016 δώσαμε 84 εκατομμύρια ευρώ σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και σε τράπεζες και σε ιδιωτικές εταιρείε. Και με μια πρώτη εκτίμηση αυτό βοήθησε στην εφαρμογή επενδυτικών προγραμμάτων περίπου 280 εκατομμυρίων ευρώ. Και όλα τα έργα αυτά τα οποία χρηματοδοτούμε δεν θα πρέπει μόνο να είναι ε, εμπορεύσουμε με τις τράπεζες, αλλά να πληρούν και αυστηρούς οικονομικούς, τεχνικούς, ε, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς όρους, γιατί πρέπει να υποστηρίξουμε πλήρως το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Το θέμα της βιωσιμότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας, βασικό για μας, γιατί είμαστε τράπεζα. Δεν είμαστε ίδρυμα παροχής επιδοτήσεων, Ούτε το θέλουμε αυτό. Ό,τι λοιπόν κάνουμε θα πρέπει να χρηματοδοτείται από τι διεθνεί αγορέ. Αν παραβιάσουμε βασικού ε, οικονομικού κανόνε, πολύ απλά οι κεφαλαγορέ, οι επενδυτέ δεν θα μα δίνουν τα χρήματα αυτά, τα 70-90 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία εκδίνει η... σε ομόλογα η τράπεζα ανά έτος. Επιπροσθέτως, και το ξέρω ότι θα σας ενδιαφέρει πολλούς από εσά. Η τράπεζά σας σήμερα εξακολουθούν όχι μόνο να είναι η τράπεζα, τα τραπεζικά ομολόγα σας είναι ε, κατεξογήν ε, πράσινα ε, ομολογά. Και δεν θέλουμε να χάσουμε σε καμία περίπτωση του επενδυτέ αυτού για τα πράσινα αυτά ομόλογα. Δεν χρειάζεται να διευκρινίσω ότι και οι τρει πυλώνε του σχεδίου Juncker είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Επικτηρωθήκαμε στο ΕΦΣΥ αλλά φυσικά θα πρέπει να βοηθήσουμε και τον κύριο Τίμερμαν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσά ω νομοθέτε, προκειμένου να παλευθούν τα προβληματικά σημεία σε ό,τι αφορά τι επενδύσει. Εδώ λοιπόν δραστηριοποιούμαστε πάρα πολύ έντονα και μαζί με την Κομισιόν και τις, έχουμε συστήσει συμβουλευτικές, ε, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την πρόθεση των έργων και την ανάπτυξη των project αυτών και για κάποιες ιδέες χρηματοδότησης. Είναι τεχνικό το θέμα και αν θέλετε θέμα τεχνικό ως προς τη χρηματοδότηση. Θα επανέλθω στο θέμα λοιπόν του αντίκτυπου της χρηματοδότησης της ΕΤΕΠ. Δεν ήθελα να μακρηγορήσω στο σημείο αυτό. Θα ήθελα να σας πω ότι είμαστε περήφανοι στην παρούσα φάση για αυτά που έχουμε πετύχει με το ΕΦΣΥ, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και βλέπουμε ότι κινούμαστε πλέον προς τις αποφάσεις για τον νέο κανονισμό και τη νέα νομοθεσία, έχουμε την ελπίδα ότι θα μας δώσετε την ευκαιρία να ε, αποκτήσουμε μεγαλύτερη εμπειρία με τις δομές διαχείρισης και δεν θα τα αναστατώσουμε πάλι όλα αυτά. Και θέλουμε επίσης ε, κριτήρια και προσωπικοποίηση των κριτηρίων. Ξέρετε για παράδειγμα ότι η απάλυνση της αλλαγής του κλίματος και η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελούν ε, από τα βασικά κριτήρια των καθημερινών μας δραστηριοτήτων. Αλλά αν θέσουμε τον πύχη τόσο ψηλά που δεν μπορούμε να τα πετύχουμε τίποτα τελικά, ουσιαστικά θα δημιουργήσουμε μια πηγή μεγάλης απογοήτευσης, κεντρικούς απογοήτευσης, γιατί πάντα θα είμαστε, θα υστερούμε σε σχέση με τις προσδοκίες. Θα θέλαμε λοιπόν να είμαστε φιλόδοξοι αλλά και ρεαλιστές. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ ε, Πρόεδρε Χόιερ. Brian Hayes από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε στην Οικονομική Επιτροπή. Είχα την ευκαιρία να σας υποδεχτώ και στην εκλογική μου περιφέρεια πριν από λίγους μήνες όταν ήρθατε για να εγκαινιάσετε το γραφείο της EIB στο Δουβλίνο και πολύ εκτιμήσαμε την παρουσία σας. Αντιμετωπίζουμε, όπως είπατε και εσείς, ένα κενό στις επενδύσεις που ξεκινά από την αρχή της κρίσης και παραμένει 600 ε, δισεκατομμύρια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξετάζοντας τις προφορίες που έχουν ε, δημοσιευτεί σχετικά με το ΕΦΣΥ μέχρι τώρα. Ορισμένε χώρες μέλη τα πάνε πολύ καλά και ιδίω εκείνε οι οποίε αντιμετώπισαν κρίσει όπω ε, αυτή που πέρασε η δική μου, δηλαδή Πορτογαλία, Ισπανία, Λιθουανία, Εστονία, Βουλγαρία. Ορισμένες από τις χώρες αυτές πέρασαν και από προγράμματα και τα κατάφεραν. Και έχουν γερό πάτημα μέσα στο ε, ε, σύστημα ΕΦΣΥ σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ τους. Τώρα, σε σύγκριση με άλλες χώρες που δεν τα πάνε τόσο καλά και σε αυτές περιλαμβάνεται και η δική μου για νέα δανειοδότηση, ποια είναι η συμβουλή σας. Είναι έλλειψη έκθεσης, το πρόβλημα έχει σχέση με τις Εθνικές Τράπεζες Πρόθεσης, έχει σχέση με τις κυβερνήσεις που ε, δεν προωθούν προτάσεις επενδύσεων σαν αυτές που θα θέλαμε να δούμε ή μήπως τελικά δεν υπάρχουν αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που να προωθούν τέτοια σχέδια επενδύσεων γιατί οπότε βλέπουμε ως τώρα η περισσότερη συμβολή για τις επενδύσεις προέρχεται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο βέβαια ανταποκρίνεται και στην εντολή που έχετε λάβει και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο. Τι συμβουλή θα δώσετε στις χώρες αυτές οι οποίες δεν προωθούν τέτοια προγράμματα. Δεύτερη ερώτηση. Γνωρίζετε ότι υπάρχει άποψη και εδώ αλλά και αλλού ότι η εντολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ίσως πρέπει να αλλάξει ώστε να μπορούν να δίνονται δανειοδοτήσεις και στην βιομηχανία εξοπλισμών. Αυτό γνωρίζω ότι θα έχει ένα ε, αντίκτυπο στην αξιοπιστία διεθνώς. Παρακαλώ το πολύ δύο λεπτά, λέει ο Πρόεδρος. Και τρία λεπτά για την απάντηση. Να με τι εννοείται κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το όριο. Νομίζω ότι οι ερωτήσεις σας απαντούν και μόνες τους περιέχουν την απάντηση. Όλα όσα είπατε είναι σωστά. Η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι κάτι που όπως είπα και πριν κανείς δεν τα σκεπτόταν αυτά το 1957. Όμως γίνεται απόλυτα κυρίαρχο το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τώρα για μας. Και δείχνει και ποιες είναι οι ελλείψεις του τραπεζικού συστήματος ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι δεν χρηματοδοτούμε ε, ανοησίες, αντίθετα Προφανώς η ανάπτυξη των δομών και το ρυθμιστικό πλαίσιο καμιά φορά για τις εμπορικές μας τράπεζες δεν είναι ευνοϊκό υπέρ της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, για μας θα παραμείνει προτεραιότητα αυτό. Δεύτερο ερώτημα που έχει σχέση με τους εταίρους μας. Όπως είπα πριν, είμαστε μια crowding in bank διότι εκδίδουμε και ομόλογα τη τάξη των 70-90 δισεκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο. Αλλά και η εμπειρία προπενταετίας όταν ήρθα εγώ στην τράπεζα ήταν ότι όταν είδαμε τι κάνει το engineering department, σε που κανένα, καμία άλλη τράπεζα δεν έχει σε όλο τον κόσμο τέτοιο πράγμα. Όταν εκδίδουμε ένα τέτοιο project, έρχονται οι ιδιώτες επενδυτές και λένε «Α, καλό πρέπει να είναι αυτό που κάνετε» και το χρηματοδοτούν. Αυτό είναι σημαντικό λοιπόν και εδώ χρειάζεται να κάνουμε προσφορές και προς τους ιδιώτες και εμπορικούς επενδυτές και στις τράπεζες, αλλά και σε εμπορικές τράπεζες. Και είναι προφανές ότι χώρες με δυναμισμό, με τράπεζες δυναμικές, εκεί αυτές αποτελούν εταίρους μας με τους οποίους μπορούμε να προχωρήσουμε σε σημαντικές επενδύσεις. Γνωρίζω ότι για παράδειγμα σε ορισμένες χώρες, Ιταλία και Ισπανία, πού θα βρισκόμασταν στις χώρες αυτές με το πρόγραμμα ΕΚΟ για παράδειγμα και άλλα. Πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία μεταξύ της Εθνικής και της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Τράπεζας. Βλέπουμε επίσης την ανάγκη ενίσχυσης Με συγχωρείτε μήπως υπερεύει το χρονικό όριο. Καλά, αφαιρέστε το χρόνο από την επόμενη απάντησή μου. Γιατί άμα αρχίσω να μιλώ για ε, υπηρεσίε παροχή συμβουλών μπορώ να σα μιλώ για πάντα. Η Περβάνς Μπερέ. Να έρθω σε αυτά που ο κύριος Χέις. Ε, ε, μια πολύ, ένα πολύ εγχείρημα το οποίο χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην περιοχή του Παρισιού. Ήταν βεβαίω εκεί ο πρόεδρος της ε, ε Δημοκρατία, δεν είσαστε εσεί ο ίδιο εκεί, Impact Creation λέγεται το πρόγραμμα αυτό ε, και προβλέπει επενδύσει σε ε, κοινωνικά δύσκολες ε, περιοχές. Εσεί πάντως συγκρίνατε την τράπεζά σα με την ικανότητα παρέμβαση της παγκόσμια τράπεζα. Ακούμε τώρα ότι η Ελλάδα, για παράδειγμα, ενδέχεται να ενδιαφέρεται για μια δανειοδότηση από την Παγκόσμια Τράπεζα. Πώς είναι δυνατόν ε, να μην έρχεται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να ζητήσει. Για μας είναι ενδιαφέρον να το γνωρίζουμε αυτό. Ε, εξάλλου, όταν εξετάζει κανείς το σχέδιο επενδύσεων Juncker μας λένε και είπατε και εσείς πόσο σημα... μεγάλη είναι η σημασία του για την αλλαγή του επενδυτικού σχεδιασμού στην Ευρώπη. Όμως, σε ό,τι αφορά τη μακρο... μακροοικονομική επίπτωση δεν έχουμε φτάσει ακόμα στα αποθούμενα αποτελέσματα και όταν βλέπω και την λίστα, δεν έχω κάνει βέβαια την πρόσθεση, λέτε ότι είναι ε, ποσά τα οποία προστίθενται ανατομέα. Αυτό που βρίσκω ότι είναι αναγκαίο ως επένδυση για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που γνωρίζουμε, τι προτείνεται ακριβώς για να πληρωθεί το κενό αυτό επενδύσεων. Απάντηση. Δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει από τον δημόσιο τομέα μόνο του και από τις δημόσιες τράπεζες μόνες τους. Εμείς προσφέρουμε βοήθεια, σημαντική νομίζω, και οι εθνικές τράπεζες κάνουν σπουδαία δουλειά, αλλά το περιβάλλον των επενδύσεων στην Ευρώπη πρέπει να βελτιωθεί. Εκεί το μεγαλύτερο βάρος φέρει νομίζω και ο Στίμερμανς και οι συναδελφοί του που προσπαθούν να καταργήσουν τις, τα, τα κολλήματα, τα εμπόδια στις επενδύσεις. Υπάρχει μια διάσταση όπου εκεί εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτικός διότι δεν είναι και της άμεσης αρμοδιότητάς μου και είναι και κάπως επικίνδυνο η επιτυχής προσπάθεια να ξεκαθαρίσει το τραπεζικό τοπίο μετά από την κρίση ενδέχεται εκεί να υπήρξαν κάποιοι τομείς όπου το παρακάναμε. Εάν εξετάσετε τις ανάγκες υποβολής αναφορών, για παράδειγμα, στις μικρές ε, επιδοτήσεις, μικρές επενδύσεις, βλέπετε ότι είναι τεράστια η υποχρέωση υποβολής αναφορών και μειώνει την ικανότητα των μικρών αυτών πιστοτικών ιδρυμάτων να χορηγούν πιστώσεις. Γι' αυτό ερχόμαστε μετά σε μεγάλες τράπεζες και ζητούμε μεγάλα ε, δάνεια για μικρόμεσες επιχειρήσεις. Για την Ελλάδα. Συνήθως θα ανέμενα η Παγκόσμια Τράπεζα ε, να ασχολείται με αναπτυσσόμενες χώρες και δεν μπορώ να πω ότι η Ελλάδα είναι αναπτυσσόμενη χώρα. Όμως αντιλαμβάνομαι την ανάγκη και χαίρομαι για την προσπάθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας. Εμείς με την έκθεσή μας στην Ελλάδα φτάνουμε το 10% του ελληνικού ΑΕΠ. Έχουμε παραμείνει εκεί και παραμείναμε στην Ελλάδα ως η μοναδική τράπεζα επενδύσεων και έχουμε φτάσει σε μια απίστευτη διάσταση εκεί και κάθε ένας που ε, συμβάλλει λοιπόν σε βοήθεια προς την Ελλάδα είναι καλοδεχούμενος για μας. Ευχαριστώ Ρόμπερτ Ζήλε. Ευχαριστώ και για την ε, περιεκτική δήλωσή σας και για τις άμεσες απαντήσεις σας. Είπατε σωστά ότι η ανάγκη επενδύσεων για χώρες συνοχής είναι προφανής και εν μέρει αυτό προσπαθείτε να κάνετε. Από την διαστρωτική άποψη, για παράδειγμα, τομέα των μεταφορών ήταν λιγότερο προφανής, λιγότερο εμφανής για σας. Βλέπουμε ωστόσο κάποιες εξελίξεις σε αυτή την τομεακή προσέγγιση. Αν δούμε όμως ποιοι είναι οι εταίροι των των ε, επενδύσεών σας. Είναι οι τοπικές κοινότητες, στην Ανατολική Ευρώπη τουλάχιστον, και βλέπουμε και ιδιωτική χρηματοδότηση, που αυτός είναι και ο στόχος βέβαια, να ενθαρρυνθεί η ιδιωτική επένδυση, διότι πώς λειτουργεί σε πολλές περιπτώσεις. Είστε ικανοποιημένο με έναν εταίρο, για παράδειγμα για την επένδυση σε έργα μεταφορών και αναμένεται οι τοπικές κοινότητες, δήμοι κλπ. να δανειοδοτηθούν από την αγορά. Το κάνουν αυτό. Αλλά τελικά αν χαθούν χρήματα είναι δημόσια χρήματα, δεν είναι ιδιωτικά χρήματα. Είναι λοιπόν επικίνδυνη η κατάσταση και ιδίω για το δημόσιο τομέα που λένε ότι πρέπει να λάβουμε μεγαλύτερη δανειοδότηση αλλά και το σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξης δεν πρέπει να επηρεάζεται από τι χρηματοδοτήσει αυτέ. Αυτό είναι υπόθεση των Υπουργών Οικονομικών. Δεν θεωρείτε κι εσείς ότι εκεί προκύπτει μια δυσκολία και πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε έτσι στα επόμενα χρόνια. Αντιλαμβάνομαι τους κινδύνους, ναι. Και αντιλαμβάνομαι και την ανάγκη, όπω πάντα στον τραπεζικό κλάδο, να διαχειριστούμε του κινδύνου αυτού. Δεν γίνεται να σφάλισουμε τα μάτια και να τα αγνοήσουμε αυτά. Πρέπει να διαχειριστούμε του κινδύνου αυτού. Και γι' αυτό λοιπόν, μαζί με του συναδέλφου από τις οικονομικές υπηρεσίε και από τη Γυροστόν θα πρέπει να καταρτήσουμε ένα εγχειρίδιο για τους Δήμου και τις περιφέρειες. Για το πώς... μπορούν να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους ευρωπαϊκούς πόρους, πρώτον, Δεύτερον, να βοηθήσουμε την ΕΤΕΠ να υποστηρίξει και κατά τρίτον να τα συνδυάσουμε αυτά με τρόπο που είναι συμβατός με το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Αυτό το εγχειρίδιο λοιπόν θα πρέπει να δημοσιευθεί. Δημοσιεύτηκε πριν από 5-6 μήνε και πραγματικά αποτελεί, έχει γίνει ενάρπαστο. Βοηθάει να ξεπεράσουμε τις αμφιβολίες για την χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων, γιατί σε πολλές χώρες ε, δεν ε, τα πιστεύει αυτά ο κόσμος, γιατί πιστεύει καταρχάς ότι είναι πολύ ακριβά. Δεν ε, είναι απαραίτητα αυτά όμως σε καμία περίπτωση και κατά δεύτερον θεωρεί ότι ευθύνονται εν μέρει για την χρηματοπιστωτική κρίση. Άρα πιστεύω ότι θα πρέπει να εξηγήσουμε καλύτερα τους τρόπους αυτούς χρηματοδότησης και την συνδυασμό του ΕΦΣΥ με το ESIF. Ελπίζω αυτό να συμβεί στο νέο κανονισμό, γιατί πιστεύω ιδιαίτερα ότι το χρειάζονται αυτό οι περιοχές που αναφέρατε. Γιατί ως τώρα τα πηγαίνουν ε, αρκετά άσχημα σε ό,τι αφορά το ΕΦΣΙ αυτές οι περιοχές. Μπορούν να βελτιώσουν πολύ τη θέση τους, θεωρώ. Ευχαριστώ, ε, κυρία Γκουλάγ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχα μια ερώτηση. Αυτή την εβδομάδα γιορτάσαμε τα 10 χρόνια του Ευρωπαϊκού ε, Συμβουλίου Έρευνας. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν με ποιο τρόπο συνδυάζουμε τα διάφορα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Βασικό χαρακτηριστικό του European Research Council είναι να δίνει μέσα με βάση την αριστεία σε Ευρωπαίους ερευνητές ε, χωρίς να κάνει αναλύσεις γεωγραφικές κτλ. Υπάρχουν βέβαια κάποιες χώρες που εξ αυτού εποφελούνται περισσότερο και πολλοί πιστεύουν ότι έτσι οι ισχυρότεροι γίνονται ακόμα ισχυρότεροι και οι ασθενέστεροι ακόμα πιο ασθενεί. Πώς μπορούμε να το ρυθμίσουμε αυτό, ιδιαίτερα στον τομέα της βασικής έρευνας, ίσως με ερευνητικά κέντρα σε πανεπιστημιακό επίπεδο, Αναφερθήκατε στα χρήματα τα οποία στρέφονται στον τομέα της ψηφιακής αγοράς και στα πλαίσια του Horizon 2020. Νομίζω ότι και το τι κάνουν τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο φυσικά είναι σημαντικό έτσι ώστε το σύνολο της Ευρώπης να προχωρήσει προς τα εμπρός. Το είπα στην αρχή ε, ότι εγώ ξέρω ότι ελέγχομαι από το διεθνή ανταγωνισμό και αυτό είναι βασικό πρόβλημα για την Ευρώπη στο μέλλον. Αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ενισχύοντας τους ισχυρούς και αφήνοντας τους φτωχούς πίσω. Όταν ταξιδεύω στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπω πολλές φορές την κατάσταση όχι μόνο των ερευνητικών ιδρυμάτων, γιατί αυτό είναι η κορυφή πολλές φορές, αλλά την ε, απαράδεκτη κατάσταση των σχολικών κτηρίων ας πούμε. Οπότε καταλαβαίνω ότι εκεί έχουμε συγκεκριμένες ευθύνες ε, για το μέλλον και για τα παιδιά της Ευρώπης. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να βρούμε τα χρήματα είτε από τα κράτη-μέλη, από τις περιφέρειες, από τις πόλεις, και να χρησιμοποιήσουμε και τον πολλαπλασιαστικό, ε, αν θέλετε, ε, την πολλαπλασιαστική μας δυνατότητα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να μιλάμε για την χρηματοδότηση μόνο των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά θα πρέπει να βελτιώσουμε το σύνολο της εκπαιδευτικής αλυσίδας από την αρχή του σχολείου μέχρι την έρευνα την πανεπιστημιακή. Βλέπω λοιπόν ότι σε πάρα πολλές χώρες υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ε, ανάγκη ε, και ιδιαίτερα σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Αν το πετύχουμε αυτό θα έχουμε κερδίσει το παιχνίδι. Επίσης θα πρέπει να αναθεωρήσουμε εν μέρη και το νομοθετικό μας περιβάλλον, γιατί η βασική μας αδυναμία είναι ότι στην βασική έρευνα και στην ανάπτυξη των έξυπνων προϊόντων μπορεί να είμαστε πρώτοι στον κόσμο σε πάρα πολλούς ε, τομείς. Αλλά αφή στιγμή οριμάσουν για την αγορά τα νέα αυτά προϊόντα, τότε έχουμε περιορισμούς με την ε, εισδοχή των προϊόντων αυτών στην αγορά. Θα πρέπει λοιπόν ε, να δούμε γιατί πλημμυρίζουμε από κορεατικά ή αμερικανικά προϊόντα σε κάποιους τομείς και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συνδέσουμε καλύτερα την φάση ανάπτυξης ενός προϊόντος και την ένταξή του στις ε, διαδικασίες των αγορών και στα πλαίσια του Horizon 2020 και με άλλες δραστηριότητες θα πρέπει να πετύχουμε πολλά, γιατί η καινοτομία δυστυχώς στις προτεραιότητες της Ένωσης δεν είναι εκεί που πρέπει. Λόπες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σας κύριε Χόγερ. Τρεις ερωτήσεις θα ήθελα να σας θέσω. Δεν ξέρω αν με βλέπετε. Λοιπόν, έχω κάποιες ερωτήσεις τις οποίες πρέπει να σας θέσω. Η πρώτη ερώτηση αναφέρεται στο ε, στρατηγικό σχέδιο επενδύσεων. Δεν θα σας ρωτήσω για τον αριθμό των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται, αλλά ε, γιατί ε, τι αναλογικότητα είναι αυτή η οποία υπάρχει. Μία βελτίωση της κατάστασης σημαίνει ότι ε, θα υπάρξει μια συνέχιση αύξηση των επενδύσεων, αλλά οι πολιτικές λιτότητας δεν το επιτρέπουν αυτό. Το στρατηγικό ε, σχέδιο αυτό δεν έχει βοηθήσει λοιπόν κάποιες χώρες, περιπλέκει αν θέλετε την χρηματοδότηση και το ίδιο ισχύει και για την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων. Μέχρι τώρα τα, τα πράγματα στον τομέα αυτό πήγαιναν σχετικά καλά στην Ισπανία. Ε, το ελεγκτικό συνέδριο σαν παράδειγμα έχει αμφιβολίες για την διεύρυνση του ΕΦΣΙ στο μέλλον για τους λόγους τους οποίους προανέφερα. Ε, στην ουσία έχουμε να κάνουμε με μια διακοσμητική αν θέλετε ε, παρουσίαση των προηγούμενων δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κάτι το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα στο ευρωπαϊκό μέλλον. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη και το θέμα της χάρτας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών συγγνώμη δικαιωμάτων. μπορείτε να μας πείτε την άποψή σας για την χάρτα αυτή και σέβεστε κάποιο πρωτόκολλο έτσι ώστε οι χρηματοδοτήσεις σας να μην πηγαίνουν ας πούμε ε, στην Σαχάρα την Δυτική ή στην Παλαιστίνη, σε κατεχόμενα ε, εδάφη δηλαδή. Εμείς ε, πολλές φορές λειτουργούμε σαν βουλευτές ως πρέσβεις ε, συγκεκριμένων προγραμμάτων. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω για τη Μούρθια στην Ισπανία, στη Λόρκα, ε, είχε ξεκινήσει από το 2011 οι προσπάθειες αδικοδόμησης της πόλης μετά από τους σεισμούς. Δυστυχώς έπρεπε να ολοκληρωθούν τα μέτρα αυτά το 2017, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα. Ο Πρόεδρος, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. κάνουμε να συνεχίσουμε. Γραπτά αν θέλετε να, κάνετε τις υπόλοιπες ερωτήσεις, αλλά δεν θα μπορούσαμε να ακούσουμε τις, απάντηση, τις απαντήσεις. Φυσικά και δεν συμφωνώ με τις αμφιβολίες που εκφράζει το ελεκτικό συνέδριο, αλλά πρέπει να τις πάρουμε σοβαρά. Και αυτό επειδή μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την συμπληρωματικότητα του ΕΦΣΥ τόσο εύκολα, γιατί κάθε έργο, είτε πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για μεγάλο εταιρικό ή δημόσιο σχέδιο, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι το μεμονωμένο αυτό ε, έργο θα μπορούσε να έχει, να έχει χρηματοδοτηθεί και χωρίς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, εννοείται. Αλλά δεν υπάρχει επίσης καμία αμφιβολία για το ότι το ΕΦΣΥ επιτρέπει στην όμιλο της ΕΤΕΠ να αυξήσει τις δραστηριότητες αυτές σημαντικά με ένα προφίλ κινδύνου το οποίο είναι πολύ πιο υψηλό σε ό,τι αφορά τις παραδοσιακές χρηματοδοτήσεις. Άρα δεν μπορούμε απλά να ισχυριστούμε ότι πρόκειται για μια επέκταση τέτοιων επενδύσεων οι οποίες θα είχαν γίνει έτσι κι αλλιώς. Δεν αληθεύει αυτό, δεν στέκει. Πριν το ΕΦΣΥ η ΕΤΕΠ μπορούσε να εκτελέσει μόνο ένα περιορισμένο ποσοστό τέτοιων επενδύσεων υψηλού κινδύνου. 6% μόνο σε σχέση με το συνολικό ποσοστό επενδύσεών μας. Και χάρη στην ευρωπαϊκή εγγύηση, τώρα 30% των υπογραφών μπορούν να συγκαταλεχθούν σε αυτές τις ιδιαίτερες αυτές ε, δραστηριότητε υψηλού κινδύνου το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων αναμένεται να αυξήσει τις επενδύσεις από 4 έως 20 δισεκατομμύρια ανά έτος. Άρα πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό από πλευράς χαρτοφυλακίου, όχι από το μεμονωμένο project, το εκάστοτε μεμονωμένο project, σε ό,τι αφορά τώρα το ερώτημα για τα τα δικαιώματα. Αυτό είναι αναπόσπαστος τμήμα της ε, έρευνας ε, για τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο κάθε έργο περνάνε όλα αυτά από πολύ αυστηρό έλεγχο και νομίζω ότι και ο μηχανισμός καταγγελίας μας και η αρμόδια ομάδα είναι πολύ αυστηρή. Προσπαθούμε λοιπόν να αφαιρούμε, να επιλύουμε ενδεχόμενα προβλήματα, συμπεριλαμβάνουμε και την διάσταση της τερικής ευθύνη. Και νομίζω ότι είναι πολύ υπεύθυνη η αντίδρασή μας, γιατί μου ήρθε τώρα πολύ απλά, δεν έχω τα στοιχεία που χρειάζονται για να σας απαντήσω, γιατί δεν γνωρίζω το συγκεκριμένο έργο, θα σας παρέχω γραπτά τις ερωτήσεις αυτές. Τις απαντήσεις αυτές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κέιτο, Σκοτ Κέιτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πέρσι η ΕΤΕΠ επένδυσε 19 δις λίρες, ευρώ μάλλον, σε ό,τι αφορά έργα για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και είπατε εισαγωγικά ότι είμαστε ηγετική δύναμη σε, τέτοια, σε τέτοιες επενδύσεις. Επειδή είναι από τους πράσινους, καλωσορίζω λοιπόν τον στόχο της ΕΤΕΠ για 20% από ανανεώσιμες μέχρι το 2020, αλλά αυτό θα σημαίνει να σταματήσουν και οι επενδύσεις σε ορεκτά καύσιμα. Ρωτώ λοιπόν, τι γίνεται στην παρούσα φάση, τι ποσοστό επενδύεται σε ορυκτά καύσιμα και πότε αναμένεται να τερματιστούν αυτέ οι επενδύσει σε ορυκτά καύσιμα. Και μία ερώτηση για το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα ξέρετε ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ιδιωτικοποιεί την δική μα πράσινη τράπεζα και ότι χρηματοδοτούν σε διάφορε περιστάσει και ορυκτά καύσιμα και όχι ανανεώσιμε. Πείτε μα λοιπόν πώ εκτιμάτε την επιτυχία του Ηνωμένου Βασιλείου για πρόσβαση σε χρηματοδότηση από το ΕΦΣΥ και από την ΕΤΕΠ ε, για τέτοια προγράμματα πράσινης οικονομίας. Πιστεύετε ότι πρόκειται για μια επιτυχία? Και τι γίνεται με το στόχο του 20% μέχρι το 2020 για τη δική μου χώρα, για το Ηνωμένο Βασίλειο. Η απάντηση σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή και τις σχετικές δραστηριότητες. Τι δράση που αναλαμβάνετε. Η τράπεζά σας είναι κορυφαία σε ό,τι αφορά τα πολυμερή χρηματοδοτικά θασμικά όργανα. Αυτό κατέστη σαφές για το G20. Ήμασταν ηγετική δύναμη στη Λίμα για την προετοιμασία λοιπόν των περιφερειακών τραπεζών από κοινού. Εμείς είμαστε ηγετική δύναμη και δείξαμε πόσο δεσμευμένοι είμαστε για το COP21. Παρουσιάσαμε στη συνέχεια σαφή στόχου, 25% χρηματοδότησης και παροχής δανείων για την μείωση της αλλαγής του κλίματος και άμεσα περάσαμε το κάθε δοκιμή τότε και υποσχεθήκαμε 35% για κάθε δραστηριότητα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάθε δραστηριότητα που έχει να κάνει με την καταπολέμηση τη αλλαγή του κλίματο. Θα το έχουμε πετύχει αυτό και μέχρι το 2020. Τώρα σε ό,τι αφορά τον Brexit. Αυτό θα αποτελέσει τεράστια απώλεια για όλου μα και ιδιαίτερα όμω για την τράπεζά μα Γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν και είναι ένα από του ισχυρότερου εταίρου μα σε ό,τι αφορά τι δράσει για την, το κλίμα και για την ενεργειακή αποδοτικότητα και για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και θα μα λείψει από τον ισολογισμό μα αυτό και από τα επιτεύγματα μας τα οποία σα παρουσιάζουμε και εσά και σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω να βρούμε έναν τρόπο να αντισταθμίσουμε την απώλεια αυτή η οποία ήταν μεγάλη η προσωπική μου άποψη σε ό,τι αφορά την πράσινη τράπεζα επειδή στο παρελθόν Ήμουν πολύ καλά ενήμερος για τα έργα αυτά και προφανώς μου προκαλεί μεγάλη λύπη το ότι θα αποχωρήσει το θεσμικό αυτό όργανο, αλλά πολύ απλά δεν μπορώ να σχολιάσω, δεν είναι δουλειά μου. Συνολικά θα μας λείψει το Ηνωμένο Βασίλειο σε ό,τι αφορά την ε, ενεργειακή αποδοτικότητα, την αλλαγή του κλίματος, αλλά και σε ό,τι αφορά την εξέλιξη. Αυτό θεωρώ ότι είναι ο κόδωνα του κινδύνου για όλου του υπόλοιπου. Αν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει σε ηγετική θέση στον τομέα αυτό, ε, θα πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια. Μάλιστα, να κάνω μια επερώτηση, μάλλον να διευκρινίσω την ερώτηση για τα ρεύτα καύσιμα. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η ενεργειακή μα πολιτική είναι ουδέτερη σε ό,τι αφορά τον τύπο ενέργειας που παράγεται. Έχουμε πολύ υψηλά πρότυπα και προδιαγραφές σε ό,τι αφορά τα όρια εκπομπών, αλλά δεν μπορούμε να προδιαγράψουμε στα κράτη-μέλη τι είδους ενέργεια θα προτιμήσουν. Αυτή τη στιγμή σκληρούνται οι όροι για τις ε, εκπομπές που είναι πολύ αυστηροί. Αν θα θέλαμε να κινηθούμε πέρα από αυτό το επίπεδο, αυτό θα έπρεπε να γίνει με πολιτική απόφαση των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Άνεμαντς. Θα μιλήσω στα Ολλανδικά, αν μου επιτρέπετε. Να σας ρωτήσω για το ρόλο τον οποίο θα αναλάβει η ΕΤΕΠ σε ό,τι αφορά την μετανάστευση και το προσφυγικό και πιο συγκεκριμένα στην πρωτοβουλία για την απεκτικότητα και στα εξωτερικά σχέδια επένδυσης αναφέρεται και αυτή η διάσταση και στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 5,3 δισεκατομμύρια έχει αυξήσει μάλλον τις εγγύσεις σε 5,3 δισεκατομμύρια και διαπιστώνουμε τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την διαφάνεια, με την ε, χρηματοδότηση, με τον έλεγχο των αυταρχικών καθεστώτων τον οποίων αντιμετωπίζετε συχνά. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι πώς κρίνετε εσείς τον νέο ρόλο τον οποίο αναλαμβάνετε από τις πολιτικές οντότητες, από τους πολιτικούς, γιατί εσείς ουσιαστικά άλλο καθήκοντα έχετε και ενδεχομένω να μην έχετε και το απαραίτητο τις απαραίτητες γνώσεις, την απαραίτητη τεχνογνωσία για να επιτελέσετε τα καθήκοντα αυτά. Πώς συγκεκριμένα θα τα καταφέρετε, πιστεύετε. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η ΕΤΕΠ δραστηριοποιείται εξ αρχής από την ίδρυσή της εκτός της Ευρωπαϊκής της Ένωσης με 10% του όγκου χρηματοδότησης, περίπου 10 δις ανά έτος. Πρόκειται για μεγάλο πόσο σε ό,τι αφορά την Αφρική για παράδειγμα. Στην παρούσα φάση είμαστε παρόντες σε όλη την Ήπειρο, γιατί έχουμε ιδιαίτερη εντολή για συνεργασία με τις χώρες ΑΚΕ. Άρα, είμαστε παρός, παρόντες εκεί. Δεν είναι άγνωστη περιοχή η Αφρική για μας, σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της ε, μεταναστευτικής ε, κρίσης, που πήρε λίγο χρόνο. Περίεργος πώς. Θυμάμαι σε μια συνεδρίαση του Συμβουλίου, όπου επεσήμανε το γεγονός ότι η ανάγκη ήταν να ανταποκριθούμε ε, προφανώς στην μεταναστευτική κρίση γιατί αυτό ε, θα προαπαιτήσει ασφαλώς χρηματοδότηση, επενδύσεις μάλλον. Και το είπα αυτό στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων τότε θα χρειαστούν επενδύσεις. Τεράστιες επενδύσεις. Και στην τελική ανάλυση αυτό στα δικά ε, τραπέζι τραπέζια θα καταλήξει. Και το θέμα το μόνο ήταν κατά πόσον θα αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα τα βαθύτερα αίτια τη κρίση. Έχει καταθέσει πλέον μια πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ευχαριστώ γι' αυτό. Αλλά σίγουρα θα μα πάρει λίγο χρόνο. Το συζητάμε εδώ και μισό χρόνο το θέμα αυτό. Δεν έχει συμβεί ακόμα τίποτε. Ελπίζω να τα ολοκληρώσει όλα αυτά λίγο η Μαλτέζικη Προεδρία. Τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, αλλά έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Η πρωτοβουλία ανθεκτικότητα ε, κατόπιν ετήματο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πριν από ένα χρόνο έχει δρομολογηθεί. Υποστηρίζω λοιπόν την πρωτοβουλία αυτή. Γιατί είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη, για την εγγύηση, αλλά χρειαζόμαστε ακόμα δισεκατομμύρια 120 δισεκατομμύρια από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το 2020 είναι μεγάλο το ποσό. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή θα ακολουθήσει και την μεταναστευτική κρίση, ας κάνουμε αυτά που πρέπει τώρα. Έχει δρομολογηθεί λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία αντακτικότητα αντοχή και θα εξασφαλίσουμε ότι κάποια στιγμή θα είναι αναπόσπαστο τμήμα του σχεδίου του επενδυτικού. Και είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι γι' αυτό. Και παρεπιπτόντω με πολύ καλή συνεργασία με άλλα πολυμερή θεσμικά όργανα και θέλουμε βασικά στην Αφρική να τονώσουμε τις δυνατότητες των ε, νεαρών επιχειρηματιών. 1.500 σε διάφορες χώρες. Θα πρέπει να αποστρεφθούν λοιπόν τα έργα αυτά και θεωρώ ότι η τράπεζα δεν προσπαθεί να αντικαταστήσει επιδοτήσεις. Όχι, προσπαθεί να δώσει οικονομική προοπτική για κάποιους οι οποίοι εξετάζουν το δεχόμενο να παραμείνουν στην πατρίδα τους. Είναι πολύ καλή προοπτική αυτή. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα πρέπει να ομαδοποιήσουμε τώρα τις ρωτήσεις. Ο κύριος Κίρτσος από την πρώτη ομάδα. Thank you, Chairman. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα Επενδύσεων είναι ένα, μια επιτυχής προσπάθεια γενικά. Πολλοί από τους συναδέλφους όμως θεωρούν ότι η τράπεζα θα μπορούσε να προωθήσει περισσότερο ένα δίκαιο φορολογικό ε, σύστημα εφαρμόζοντας τους κανόνες με τους ενδιαμέσους με τους οποίους συνεργάζεται. Θα μπορούσατε να τους πείσετε να υιοθετήσουν σωστούς κανόνες ή θα πρέπει η εθνική νομοθεσία ε, να προσαρμόζεται στα συμφέροντα των ενδιαμέσων. Έχω και μια δεύτερη ερώτηση. Μπορείτε να μας πείτε κάποια επιπλέον στοιχεία για την κατάσταση στο Brexit και την τράπεζά σας. Υπάρχουν πολλά προγράμματα στα οποία εμπλέκεται το Ηνωμένο Βασίλειο. Πώς θα αλλάξει η ζωή σας μετά το Brexit. Συλλέγουμε ερωτήσεις προς το παρόν. Ιβάν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να θέσω μια πάρα πολύ σύντομη ερώτηση η οποία σχετίζεται με ένας από τους βασικούς στόχους της τράπεζας, την κινητοποίηση των επενδύσεων δηλαδή στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε αναπτυγμένες ε, οικονομίες ε, όπου υπάρχουν επενδύσεις, όπου υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη, όπου υπάρχει παράδοση θα έλεγα για την εφαρμογή μεγάλων προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών μίξ από πολλαπλές πηγές. Όμως ταυτόχρονα υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες οι οποίες υποφέρουν από το λεγόμενο χρηματοδοτικό κενό και σε αυτές τις χώρες υπάρχουν και κάποιες ε, περιοχές όχι πολύ αναπτυγμένες, οι οποίες δεν έχουν ούτε την εμπειρογνωμοσύνη, ούτε την, θα έλεγα, παράδοση διαχείρισης τέτοιων προγραμμάτων. Θα πρέπει λοιπόν η τράπεζά σας να λαμβάνει υπόψη και κάποια επιτέλους γεωγραφικά κριτήρια, έτσι ώστε οι επενδύσεις να κατανεμηθούν δικαίως, ε, ισότιμα και η τράπεζά σας μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέχει τις εμπειρίες και τις συμβουλές οι οποίες απαιτούνται και αναφέρομαι εδώ σε κομμάτια της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Thank you, uh, Mr. Mato. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Νομίζω ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκουν μια μεγαλύτερη προσθετικότητα. Οι προτάσεις γενικά πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα ήθελα να μην μείνει η προσθετικότητα σε θεωρητικό επίπεδο, θέλω να χαρακτηρίζει τα μεμονωμένα προγράμματα. Και τώρα για την εμπλοκή των εθνικών τραπεζών επενδύσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, θα πρέπει να γίνουν πιο φιλόδοξες αυτές ε, οι τράπεζες σε εθνικό επίπεδο. Ποια είναι η γνώμη σας γύρω από αυτό και εσείς είστε διατεθειμένος να συνεργαστείτε με πιο συντονισμένο τρόπο με αυτές τις τράπεζες. Μπορείτε να απαντήσετε λέει ο πρόεδρος τον κύριο Χόγερ. Για τον κύριο Κίρτσο θέλω να σας ευχαριστήσω για την στήριξή σας και την συνεργασία σας και για τις βαθύτατες γνώσεις που έχετε γύρω από το ε, όργανο το δικό μας. Για την συγκεκριμένη ερώτηση τώρα την οποία θέσατε, για την προώθηση ενός δικαίου και διαφανούς φορολογικού συστήματος και σε ποιο βαθμό μπορούμε να το πετύχουμε και μέσω των συμβατικών μας ε, υποχρεώσεων. Ε, Εμεί παίρνουμε μέρος στα Global Forum για την ε, διαφάνεια στη φορολογία και θέλουμε να προωθηθεί ένα τέτοιο σύστημα. Η τράπεζα παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε τα επίπεδα τα δικά μας να είναι συμβατά με τις διεθνείς εκτελήξεις. Οι βέλτιστες πιστοτικές πρακτικές σαν παράδειγμα λαμβάνονται υπόψη και όταν γίνονται αλλαγές και ρυθμίσεις στα φορολογικά συστήματα παίρνουμε μέτρα έτσι ώστε να βελτιώσουμε την συνειδητοποίηση και τον έλεγχο που έχουμε των αλλαγών αυτών για να συνεισφέρουμε στην καταπολέμηση των, φορο, των μορφών φοροδιαφυγής. Και τα προγράμματά μας στα πλαίσια της λεγόμενης πρακτικής της due diligence προσπαθούν να ανταποκρίνονται σε αυτό το οποίο είπατε. Θα πρέπει όμως να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να συμμετέχουμε σε όλα τα διεθνή φόρα τα οποία ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα για το Brexit, ε, ε, χάλια θα είναι η ζωή μας, χάλια, χάλια όταν φύγουν οι Άγγλοι. Ε, και στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι άσχημη η κατάσταση, αλλά έτσι είναι τα πράγματα και λυπάμαι βαθύτατα για αυτό που θα συμβεί. Εγώ συζήτησα με τον Πρόεδρο πριν συναντηθούμε εδώ ανεπίσημα ότι θα πρέπει η ομάδα του Κοινοβουλίου που ασχολείται με τις διαπραγματεύσεις να σχηματίσουμε μια πλήρη εικόνα της σημασίας της Τράπεζας Επενδύσεων δεν είναι θέμα αριθμών μόνο και αμοιβαίων διεκδικήσεων, δεν είναι εκεί το θέμα, αυτό θα ήταν ε, πραγματικά παράδεκτο. Το θέμα είναι να δούμε ε, ε, ποιο ρόλο παίζει η τράπεζά μας στα πλαίσια του Brexit. Και αυτό είναι σημαντικό και για τον ίδιο τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Βέβαια η EIB δεν είναι τμήμα του προϋπολογισμού, βασίζεται στις χρηματαγορές με ε, με πραγματικά συνολικό κύκλο θα έλεγα που φτάνει τα 3-3. Ε, συγγνώμη το μισό συγγνωμη το ε, μισο 3 πραγματικα αν το συγκρίνετε ε, με αυτά τα οποία κάνουμε θα δείτε ότι το 16% των μετοχών μας ελέγχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και θα πρέπει να βρεθούν λύσεις εδώ. Θα πρέπει οι πολιτικοί ηγέτες και εσείς να έχετε την πλήρη εικόνα. Τα θέματα αυτά φυσικά είναι και ιδιαίτερα ευαίσθητα για τις χρηματαγορές, γιατί λειτουργούμε στις παγκόσμιες χρηματαγορές. Γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση και να σας δώσουμε την δυνατότητα να δείτε το πώς θα πάνε τα πράγματα. Έχουμε δημιουργήσει μια ειδική ομάδα για το Brexit, έχουμε νομομαθείς, εμπειρογνώμονες, μια ειδική λοιπόν ομάδα ιδιαίτερα έμπειρους ε, δικηγόρους, στατιστικούς που θα μας βοηθήσουν νομίζω σε μια διαδικασία οδυνηρή και απαιτητική και θα παρακολουθήσετε και εσείς τη διαδικασία Evans. Εγώ συνειδητοποιώ ποιο είναι το πρόβλημα, αλλά το ΕΦΣΙ, το στρατηγικό σχέδιο, μας δείχνει ότι κάποια αντικυκλική περιφερειακή εκπροσώπηση είναι εφικτή. Άμα βλέπετε ποιες είναι οι χώρες που έχουν ωφεληθεί περισσότερο, με την εξαίρεση της Ιταλίας και της Ισπανίας, που είναι έβδομες η ένατη, ε, είναι πολλές οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Είμαστε επιτυχείς εκεί, αλλά πολλά ακόμα μένει να γίνουν και αυτό απαιτεί την δημιουργία δυνατοτήτων και από πλευράς εθνικής. Η δική σας χώρα ιδιαίτερα νομίζω ότι η μη χρησιμοποιημένη πόρη για την προώθηση των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ ε, υψηλή και θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερα στοιχεία τον επόμενο μήνα παρέχοντας περισσότερες συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τη χώρα σας. Αλλά αν δείτε στο παρελθόν, ε, ένας από τους, ε, ε, ένα, μία από τις πιο σημαντικές νομικές υπηρεσίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι στο Βουκουρέστι. Δεν είναι κάτι που μας εκπλήσει δηλαδή, Απλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί η δυνατότητα αυτή με τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συμμετοχή των εθνικών τραπεζών για επενδύσεις και προώθηση επενδύσεων, όπως ζήτησε και ο κύριος Μάτο. Η δική σας χώρα σε σχέση με την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων είναι σημαντικό, θα έλεγα Η συνεργασία με την αρμόδια τράπεζα στην Ισπανία είναι πάρα πολύ στενή και θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Έχουμε προσφορές πολύ σημαντικές, κάνουμε και εμείς προσφορές στις αναπτυξιακές υπηρεσίες και θα πρέπει να πω ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να έχουμε συνολικά υπόψη σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η παρουσία των εθνικών επενδυτικών τραπεζών διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα. Θα πρέπει λοιπόν στο τέλος της διαδικασίας να μην είναι μόνο οι πέντε μεγαλύτερες χώρες που παίρνουν το μεγαλύτερο ποσό. Θα πρέπει να είμαστε παρόντες και σε διαφορετικές χώρες και σε χώρες που δεν υπάρχουν οι επενδυτικές τράπεζες ε, θα συνεργαστούμε με όλες τις ενδιάμεσες αυτές ε, φάσεις, στάδια, αλλά χρειάζεται η συνεργασία των διαφόρων χωρών μελών. Φερνάντες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις συγκεκριμένες. Ελπίζω να μου απαντήσετε. Το ΕΦΣΙ στην αρχή του, του στρατηγικού προγράμματος ε, Γιούνκερ Μιλήσαμε ε, για την προοπτική βελτίωση των, ε, της χρηματοδότησης αλλά και τις επενδύσεις προς τον δημόσιο τομέα. Βλέποντας λοιπόν τώρα την συμμετοχή του δημοσίου τομέα ε, και μέσω της πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί, είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στα πλαίσια του υπολογισμού και των προγραμμάτων του Darle cuál eh, la valoración que hace el BEI του eh, σύμφωνο του οικονομικού και ε, για την ανάπτυξη που ισχύει. Ε, η αλήθεια είναι ότι οι πλατφόρμες αυτές λειτουργούν περισσότερο σε κάποιες χώρες και γι' αυτό θα πρέπει να βελτιωθεί η ευελιξία αυτής της πλατφόρμας. Θα θέλαμε περισσότερα στοιχεία γι' αυτό. Μια δεύτερη ερώτηση είναι ακριβώς τα λεγόμενα συμβουλευτικά αυτά κέντρα, οι συμβουλευτικές πλατφόρμες. Αυτές είναι απαραίτητες για να βοηθήσουν και την παρουσίαση προγραμμάτων που θα διεκδικήσουν χρήματα από το πρόγραμμα Juncker. Αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν γνωρίζουμε αυτή η συμβουλευτική διαδικασία αν λειτουργεί μέχρι τώρα σωστά. Ε, ποια είναι τα προγράμματα τα οποία χρησιμοποιούν τα hubs και τα προγράμματα τα οποία ζητούν μόνα τους χρηματοδότηση. Σύγκριση δηλαδή ανάμεσα στις πλατφόρμες από τη μία και τα advisory hubs από την άλλη. Μάννα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Χόιερ. Μιλήσατε πριν για... Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Για την στήριξη πολλών μικρών και μεσών επιχειρήσεων. Θα ήθελα να φέρω και ένα άλλο παράδειγμα στην πόλη Frankfurt am Main, στο κρατήριο της Έσης. Δώσατε επίστοση πολλών εκατομμυρίων ευρώ για να οικοδομηθεί το νέο Terminal 3 του αεροδρομίου. Αναμένουμε πρόσθετους 10 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο. Σημαντικό μέτρο λοιπόν για την βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου αυτού όπου εγκαθίσταται η επιχείρηση. Υπάρχουν άλλε συνεργασίε πάλι σε αυτό το πλαίσιο μεγέθου, ας πούμε που θεωρείται ότι έχουν μια μελλοντική προοπτική διότι βεβαίω δεν είναι πάντοτε έτσι, δεν είναι άμεσα αναγνώσιμη πάντα η μελλοντική προοπτική σε όλα τα επενδυτικά σχέδια. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχεδιασμού Επενδύσεων. Σημαντικό για να γνωρίζουν οι επενδυτέ καλύτερα τι κάνουν με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντο, αλλά και οι αρχέ για παράδειγμα, ποια τεχνική υποστήριξη μπορούν να χορηγήσουν, για παράδειγμα, και σε τοπικού ενδιαφέροντος επενδυτικά εγχείρηματα, το νέο αυτό εργαλείο, το οποίο θα έχει και κάποια καινοτόμα στοιχεία, δηλαδή μια πλατφόρμα η οποία επιτρέπει χορήγηση συμβουλών και για ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν ποιες ελπίδες έχετε από αυτήν την τροποποιημένη ε, μάλλον το τροποποιημένο εργαλείο. Νίνα Γκίλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Χόιερ, συμφωνώ με τα όσα συναισθάνεστε για το Brexit. Και το πρώτο θέμα είναι ακριβώς το Brexit. Στην εκλογική μου περιφέρεια έχουμε ένα μεγάλο νοσοκομείο, το Birmingham Middle, σημαντικό έργο, το οποίο έχει ενταχθεί στους στόχους FC1. Και προσφέρει υπηρεσίες και σε έναν πληθυσμό που μεγαλώνει διαρκώς, αλλά και σε μια αναζωγόνηση ολόκληρης της περιοχής. Ποιες διασφαλίσεις μπορείτε να δώσετε και σε μένα και σε άλλους ό,τι αφορά το ότι αυτά τα σχέδια που αρχίζουν θα ολοκληρωθούν. Δεύτερο, για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ε, σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές δράσεις που θα έχετε όλο και μεγαλύτερο ρόλο για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών και προσφυγικών κρίσεων στην άμεση γειτονία της Ευρώπης με το External Investment Plan που είναι στην πραγματικότητα μια παραλλαγή του ΕΦΣΥ. Ποια διδάγματα έχετε από την ε, λειτουργία του ΕΦΣΥ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και στο EIP. Και αντιλαμβάνομαι ότι η εντολή σας για εξωτερική δανειοδότηση αναθεωρείται και ενδέχεται να υπάρξουν περικοπές σε ορισμένους τομείς όπως της Ασίας. Η ανησυχία μου είναι ορισμένα έργα τα οποία έχουν σχέση με την προσθέση του κλίματος. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αν σταματήσουν τα εγχειρήματα αυτά και για την Ευρώπη αλλά και για τις περιοχές αυτές. Και τέλος πάλι κλιματική αλλαγή θα έρθετε πάλι σε αυτό που είπε η κυρία Κέιτο. Μια από τις ανησυχίες μου είναι πώς διασφαλίζεται ότι οι επενδύσεις για την αντιμετώπιση των στόχων COP21 δεν είναι greenwashing. Τι κάνετε για να εξασφαλίσετε ότι το εργαλείο ΕΦΣΥ παίζει σημαντικό ρόλο για την επίτευξη ορισμένων στόχων που έχουμε βάλει με την διάσκεψη COP21. Κύριε Κόμπορα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς ήμουν απόν πριν. Το άρθρο 308 της Συνθήκης Λειτουργίας, μάλλον της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, απαιτεί η μέτοχοι της τράπεζας να είναι χωρισμένοι. Από τα όσα είπατε πριν, είμαι βέβαιος ότι δεν θα εκπλαγείτε να ακούσετε ότι η ε, Βρετανία θα ζητήσει πίσω τις επενδύσεις της. Ποια, είναι, ποια σχέδια κάνετε για να αντιμετωπίσετε το ενδεχόμενο αυτό. Θα τα κατανείμετε στους υπόλοιπους συμμετόχους, τα βάρια αυτά. Ή θα προσαρμόσετε το χαρτοφυλάκιό σας για να επιστρέψετε ένα μεγάλο ε, αποθεματικό σε μετρητά. Ή θα κάνετε κάποια κατανομή σε είδος για να τα επιστρέψετε αυτά στην Βρετανική κυβέρνηση. Και μήπως είναι ευκολότερο να επιτευχθούν αυτά εάν το Ηνωμένο Βασίλειο φτιάξει ένα sovereign fund για τον σκοπό αυτό. Και ποιο θεωρείτε ότι είναι εύλογο χρονικό περιθώριο για να ανταποκριθείτε στις απαιτήσει του Ηνωμένου Βασιλείου. Ευχαριστώ, λέει ο να αρχίσω με τις δραστηριότητες παροχής συμβουλών και την πλατφόρμα που νομίζω ότι έχουν κρίσιμο χαρακτήρα και μελλοντικέ εξελίξεις ε, ε, ε, είναι, είναι ενδεχόμενο να υπάρξουν και εξελίξεις και θα πρέπει να επιδιωχθούν. Θα προσφέρουμε το μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας διότι οι εταίροι μας δεν έχουν άμεση πρόσβαση στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Άρα ε, θα πρέπει να βοηθήσουμε εμείς που έχουμε. Η παροχή συμβουλών είναι κέριο χαρακτήρα και ενισχύει ιδίω τις ικανότητες των διαχειριστικών αρχών για την ανάπτυξη έργων και την εφαρμογή τους. Και αυτή είναι μια σημαντική αδυναμία σε ορισμένες χώρες της ε, νοτιο Ανατολική Ευρώπης. Οφείλουμε να το πούμε αυτό καθαρά. Είναι ένα μέγα θέμα. Για τον κύριο Φερνάντες. Financial Promotion Banks. Έχουμε 16 τέτοιε εθνικές promotion banks και θα πρέπει να δείτε ότι δεν μιλούμε μονάχα για την τράπεζα αλλά και για τη θηγατρική. Αυτό που χρειάζεται σε πολλές χώρες είναι η ενθάρρυνση του επιχειρήν για νεοφυείς επιχειρήσεις, για ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αρχίζουν τις δραστηριότητες τους και νομίζω ότι είμαστε καλά εξοπλισμένοι με το ΕΦΣΥ που δραστηριοποιείται όλο και περισσότερο σε χώρες μέλη όπου δεν ήταν παρόν πριν από δύο χρόνια και λειτουργεί καλά. Τι μου σημειώνεται εδώ. το Broadband Fund. Ε, είναι επίσης μια δυνατότητα για τις χώρες αυτές και ε, είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τα τοπικά έργα. Καμιά φορά είναι πολύ ενθαρρυντικά, πολύ, πολύ ενθαρρυντικά και άλλοτε είναι αποθαρρυντικά. Στη χώρα που γνωρίζουμε καλύτερα και εσείς και εγώ έχουμε και πολύ καλά παραδείγματα και ορισμένα πραγματικά τρομακτικά σε ό,τι αφορά τα αεροδρόμια, εννοεί τη Γερμανία. Εάν λοιπόν ένα έργο όπως αυτό στην Φραγκφούρτη αποτελεί μέρος ενός σχεδιασμού για τα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι καλό να εξετάσουμε εμεί το ενδεχόμενο επένδυση και, και με μεγάλη ικανοποίηση το κάνουμε. Όμως, άλλωστε στο παρελθόν η τράπεζα ήταν παρούσα σε, πολλά, σε πολλές ε, ε, επενδύσεις σε αεροδρόμια στην Ένωση, και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε εάν μπορούμε να προσφέρουμε τον τρόπο αυτό ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στο έργο. Και αυτό συμβαίνει εδώ. Οι προσδοκίες μου είναι σημαντικές για περαιτέρω εξέλιξη. Κάνουμε άλλωστε πολύ περισσότερα από αυτά που σημειώνουν καν τα Υπουργεία Οικονομικών ε, ότι γίνονται δηλαδή σε σχέση με τις τοπικές κοινότητες, δήμους κλπ. Και στα πλαίσια αυτά, το βιβλίο που ανέφερα πριν που εκδίδουμε μαζί με την Ευρωστάτ είναι πολύ χρήσιμο διότι καμιά φορά υπάρχει έλλειψη πρόσβαση στη γνώση σε ό,τι αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και οφείλουμε να καταβάλουμε προσπάθεια να ξεπεράσουμε κάποιες προκαταλήψεις απέναντι στα EPP για παράδειγμα. Εφόσον τα έργα χρηματοδοτούνται με νυφάλιο και καθαρό τρόπο έχουμε τόσες αρνητικές εμπειρίες από την ε, σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο παρελθόν που μπορεί ε, να αποθαρρυνθούμε. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και καλά παραδείγματα. Μία από τις καλύτερες εμπειρίες μου ήταν το Birmingham. Μου μιλήσατε για το νοσοκομείο. Αφήνω τι είπαν μετά η επικεφαλής του νοσοκομείου για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Συνολικά πάντως το εγχείρημα ήταν όρθο, ήταν θετικό και περιλαμβάνεται στις συζητήσεις που κάνουμε τώρα μεταξύ των 27 και των 28 και το μόνο που ελπίζω είναι το Brexit και απαντώ έτσι και στην τελευταία ερώτηση. Ελπίζω να φτάσουμε σε ένα πολιτισμένο τρόπο να διαπραγματευτούμε την έξοδο του, Ηνωμένου Βασιλείου, γιατί κανείς δεν έχει συμφέρον ούτε οι ασθενείς του νοσοκομείου σας, ούτε οι Πολωνέζοι νοσοκόμες που εργάζονται εκεί. Από όποια άποψη και να το κοιτάξετε το πράγμα, πρέπει να το διαπραγματευτούμε με κατάλληλο τρόπο το Brexit. Και θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση που μας περιμένει. Στα πλαίσια αυτά, η συνέχιση των δραστηριοτήτων μας στο Ηνωμένο Βασίλειο βεβαίω είναι σημαντική. Είναι μέτοχος του Ηνωμένο για την ώρα και εκτελούμε έργα, χρηματοδοτούμε έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχουν μάλιστα και πολύ καλή απήχηση στον ισολογισμό μας και δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα σταματήσουμε ή να τα διακόψουμε. Από την άλλη μεριά οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι για την ώρα το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ε, μέρο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ε, εκεί ε, ισχύει το πρωτόκολλο περί Θα δούμε τι θα γίνει όταν θα υπάρξει το Brexit δεν θα ηγούμε εγώ των διαπραγματεύσεων Brexit στα μάτια του κοινού. Θα χρειαστεί μια τεράστια προσπάθεια με τους επικεφαλείς Μπαρνιέ και Φεγόστατ. Θα προσπαθήσουμε να τους στηρίξουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Αλλά οι διαστάσεις για τις οποίες μιλούμε είναι γιγάντιες και θα χρειαστούν κάποιες ισορροπίες και είναι δύσκολο να φτάσουμε σε συμπεράσματα. Δεν είναι μονάχα το τεράστιο σύνολο περιφερειακών στοιχείων η Βρετανία έχει και 16% των μετόχων, των μετοχών συγγνώμη, και θα ζητήσει το αντίτιμο των μετοχών αυτών. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και, ε, υπάρχει και το παθητικό στο οποίο συμμετέχει επίσης η ε, Μεγάλη Βρετανία με 16% ελπίζω και εκφράζω ξανά την ελπίδα μου ότι θα μπορέσουν να διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις με το αναγκαίο πνεύμα εάν θέλουμε να συνεργαστούμε θετικά με το Ηνωμένο Βασίλειο διότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει στον χάρτη και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις περισσότερες από τις χώρες μέλη. Τώρα για το λεγόμενο greenwashing. Αυτό που είναι σημαντικό για τα project της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι ότι αυτή τη στιγμή εγκριθεί η χρηματοδότηση δεν σταματάει το έργο. Συνεχίζουμε, παρακολουθούμε το έργο μέχρι να αποπληρωθεί πλήρως. Γι' αυτό και ενδιαφερόμαστε, για παράδειγμα, στο, ε, για το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το 2052, όταν θα ολοκληρωθεί το τελευταίο έργο που χρηματοδοτούμε εκεί και θα αποπληρωθεί δηλαδή. Και αυτό είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι επενδυτές και οι project promoters εμένουν στους στόχους τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, κάθε ημέρα μετά από την, ε, ε μάλλον ε, συνεχώς και μετά από την ημέρα της υπογραφής. Γιατί υπάρχουν συμβατικές προβλέψεις ότι εάν δεν ε, γίνει αυτό μπορεί να αναζητηθεί το δάνειο. Κάλυψα όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Να με συμπαθάτε που ξεπέρασα το χρόνο, αλλά ήθελα να απαντήσω με πλήρη τρόπο στις ερωτήσεις σας. Μόνο κατά πέντε λεπτά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ε, ενδιαφέρουσα η συζήτηση και χρήσιμη όπως πάντα. Να σας ε, διαβεβαιώσω ότι το Κοινοβούλιο αντιλαμβάνεται πλήρω τη σημασία των θεμάτων που άπτονται τη ΕΤΕΠ και των διαπραγματεύσεων το, για το Brexit. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είναι θετικό ο ρόλο που θα δραματίσουμε στη διαδικασία αυτή και θα είμαστε σε στενή επαφή μαζί σα και με την τράπεζα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο Χόιερ και πλήξη της συνεδρίασης ξαναξεκινάμε στις 3.